Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Δεν έχουμε δανέζικα, φιλανδικά, σουηδικά, λετονικά, σλοβενικά, μαλτέζικα, βουλγάρικα, τσεχικά, σλοβακικά και εστονικά. Δεν έχουμε. Σήμερα το αναφέρω για να μην προκύψουν παρανόησεις. Η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται ζωντανά σε webstream. Όπως είχαμε συμφωνήσει, για την σημερινή απογευματινή συνάντηση θα αφιερώσουμε το χρόνο μας σε μια ακρόαση για τη μη διάδοση. Αύριο μπορώ να σας ανακοινώσω ότι οι εργασίες μας θα αφορούν μια συνάντηση με την κυρία Καμή Μοσάρ και μετά θα συναντήσουμε τον κύριο Αλεξάνδρ Βέης, τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης. Σήμερα, όπως είχαμε συμφωνήσει, θα αφιεράσουμε λοιπόν τις σημερινές μας εργασίες στην ακρόαση με θέμα τη μη διάδοση. Ζητήσαμε από πέντε εμπειρογνώμονες να έρθουν, τον κύριο Πασκάλ Ζαντέρς από το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας, τον κύριο Μεγέρ, τον εκπρόσωπο της Ένωσης για τον Ένοχο των Όπλων, την κυρία Καμίγ Γκρό, Διευθύντρια στο Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας στο Παρίσι, την κυρία Ρεμπέκα Τζόνσον, από το Akron Institute for Disarmament Diplomacy του Λονδίνου, και τον κύριο δόκτορα Κάρλο Μασάλα από τη στρατιωτική ακοδημία του Μονάχου. Θα δώσω το λόγο λοιπόν σε αυτούς τους πέντε εμπειρογράμμονες για 15 λεπτά της ώρας στον καθένα και μετά θα έχουμε μια συζήτηση με τα παρόντα μέλη επί του θέματος, επί των τριών, να το πω καλύτερα, βασικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ζάντες και ο κύριος Μάγερ θα μας μιλήσουν για τις νέες προοπτικές του καθεστώτος μη διάδοση εν της διάσκεψης για να θεωρήσει της NPT. Ο κύριος Καμίγι θα μας ε, αναφέρει τα των δύο ε, βασικών διεθνών κρίσεων ε, εις ό,τι αφορά τη διάδοση των όπλων Βόρεια Κορέα και Ιράν και μετά με τον κύριο Μασάλα θα ασχοληθούμε με το θέμα ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα και με τις πρόσφατες προτάσεις ε, Ομπάμα. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζάντερς και μετά στον κύριο Μάγερ. Παρακαλώ κύριε Ζάντερς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είμαι ερευνητή στο Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά θα σας παρουσιάσω τα δικά μου πορίσματα. Το λέω αυτό διότι δεν αντανακλούν αναγκαστικά τη θέση της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι Υπάρχει και μια μικρή ομάδα εργασίας στο Ινστιτούτο που εξετάζει το θέμα του μέλλοντος ε, της μη διάδοση των όπλων. Εγώ μιλώ ως μέλος αυτής της ε, ομάδος, οπότε είναι μια ευτυχής σύμπτωση. Θα είμαι σύντομο. Έχω παρουσιάσει, έχω ετοιμάσει καλύτερα μια παρουσίαση, την οποία απέστειλα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στου ε, συμμετέχοντες. Η NPT από όλε τι συμβάσει είναι αυτή που έχει τα περισσότερα μέλη. 189 κράτη από τα 194 ανεξάρτητα κράτη του κόσμου. Θα μπορούσα εδώ να προσθέσω και την Ταϊβάν. Υπάρχουν βεβαίως Ινδία, το Ισραήλ και το Πακιστάν. Και η Βόρεια Κορέα, η οποία όμως απεχώρησε στις 10 Απριλίου. Και υπάρχουν και άλλα κράτη που τελούν υπό αναγνώριση όπως το Κόσοβο. Right, and one of them is the nuclear weapon states. These are, of course, the five, equally the five permanent members of the UN. Λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ορίσει ε, τα πυρηνικά όπλα ε, ως ε, αντικείμενο αυτής της σύμβασης. Η Βόρεια Κορέα, η Ινδία και το Πακιστάν έχουν κάποια όπλα πυρηνικά, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς ποια και πόσα, επί τη βάση των δοκιμών, των πυρηνικών δοκιμών που έχουν κάνει το Ισραήλ. Είναι βεβαίως επίσης μια τέτοια περίπτωση, χώρα για την οποία πιστεύουμε, εικάζουμε ότι έχει μεγάλο πυρηνικό οπλοστάσιο. Τώρα, για το NPT ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος. Το υλικό στο οποίο βασίζονται οι χώρες για να αναπτύξουν την πυρηνική τους ικανότητα πέρα από τις γνώσεις, την τεχνική και τον εξοπλισμό, είναι όλο ένα και πιο προσβάσιμο. Και γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα μετέπειτα απόκτησης αυτού του υλικού. Αυτό το οποίο ανησυχεί είναι οι χώρες που ρητά έχουν πει στην IEA ότι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς πολύ συχνά βρίσκονται σε ασταθείς περιοχές του κόσμου όπου, που επαπειλούνται με συγκρούσεις. Η απόκτηση λοιπόν ενός ε, ακόμα και μη στρατιωτικού προγράμματος μπορεί να είναι λόγος ανησυχίας. Άλλος λόγος ανησυχίας είναι βεβαίως το γεγονός ότι όσο περισσότερα κράτη αποκτούν την σχετική τεχνολογία μπορούν να αποτελέσουν πηγή ή κόμβο μεταφοράς όπλων. όπως έγινε με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της γυντνίασής τους με χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα. Ακόμα και, όταν όμως όλα πάνε καλά, ούτως υπήν, ο μεγάλος αριθμός χωρών που αποκτούν όχι πυρηνικά όπλα, αλλά πυρηνική ικανότητα κατασκευής όπλων, τίθεται το ερώτημα αν η IAEA υπό τον ε, παρόντα της σχηματισμό μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο της εξακρίβωσης της κατάστασης και του ελέγχου των ε, εγκαταστάσεων αυτών. Μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη είναι ότι η πυρηνική συνεργασία για μη στρατιωτικούς λόγους λαμβάνει χώρα μεταξύ μη μελών της NPT που όμως ε, ε, είναι γνωστό ότι έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά όπλα. Με τις τεχνολογικές μεταφορές που ανέφερα προηγουμένως υπάρχει πρόβλημα με το Ιράν και σε λιγότερο βαθμό με το Πακιστάν και βεβαίως ορισμένες από τις βασικές αρχές ε, της συνθήκης NPT τίθενται σε αμφισβήτηση. Τέλος, αν ε, κοιτάξει κανείς ε, τις τρεις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα και που ανέφερα στην προηγούμενη διαφάνεια, θα διαπιστώσουμε ότι και οι τρεις πλήττονται από πολιτική αστάθεια. Με πιο οξία περίπτωση αυτή του Πακιστάν κατά πάσα πιθανότητα. Εντός του πλαισίου λοιπόν του NPT κατά την απόψή μου, ε, αναφύεται μια σαφής τάση ότι τα διάφορα κράτη έχουν διαφορετικό καθεστώς εντός της συνθήκης. Λόγω των διακρατικών ή ακόμα και πολλές φορές διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό αποτελεί βαθμό, ε, μάλλον λόγο ανησυχίας και πολλές χώρες διερωτώνται γιατί δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε πυρηνική τεχνολογία λόγω αυτού. Εν είδη πρόκλησης θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα που βλέπετε στην διαφάνεια. Κινούμεθα προς ένα στάδιο το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε στάδιο μη διάδοσης. Με τα χημικά και βιολογικά όπλα η απάντηση είναι ναι. Η τεχνολογία έχει εξαπλωθεί, είναι παρούσα παντού, όλοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, υπάρχουν πολλές πηγές τεχνολογίας, Δηλαδή, πολλές από τις βασικές αρχές της ε, πολιτικής μη δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή των βιολογικών και χημικών όπλων για την πυρηνική τεχνολογία. Τώρα, θα έλεγα ότι μπορεί να εισέρχεται σιγά σιγά σε αυτήν την ε, α, φάση. Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί βεβαίω θα πρέπει να ενισχύσουν την μη διάδοση, αλλά έχουν φτάσει στα ωριά του Η περίπτωση του Ιράν, α πούμε, που θα εξετάσουν πιο λεπτομέρο ο κύριος Γκροντ, Γκροντ για την ακρίβεια. Οι κυρώσεις ε, είναι τελικά αντιπαραγωγικές εις ό,τι αφορά την εξέβρεση λύσης. Διότι αυτό που γίνεται είναι ότι στην ίδια τη χώρα, παρά τις αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σύστημα, κανείς δεν τάσεται κατά της απόκτησης πυρηνικής τεχνολογίας. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να παίξει το χαρτί της πολιτικής ας πούμε ισορροπίας για να αποθαρρύνει κάποιο κομμάτι της ηθήνουσας τάξης ή του λαού να αποποιηθεί του δικαιώματος αυτού. Και βεβαίως εύκολα δικαιολογείται ε, η απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας, όπως είδαμε και με τη Βόρεια Κορέα, αλλά και με το Ιράν περίπου και σχεδόν. Τα μέσα ελέγχου λοιπόν της διάδοσης των πυρηνικών όπλων έχουν αλλάξει και είναι λιγότερο αποτελεσματικά. Ένα δεύτερο στοιχείο που θεωρώ προβληματικό είναι ότι για να γίνει η παλήθευση της κατάστασης είναι απαραίτητη η συνεργασία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Με τις επιθεωρήσεις, όπου η χώρα δεν μπορεί να αρνηθεί τις επιθεωρήσεις αυτές κτλ. Εδώ υπάρχει μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων πριν οι επιθεωρητές λάβουν το πράσινο φως για να εισέλθουν στην ε, χώρα για να διενεργήσουν τους ελέγχους. Και βεβαίως το θέμα είναι άκρος πολιτικό, όχι μόνο στην ε, IEA, και το διοικητικό της ε, όργανο, συμβούλιο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν είναι και αυτές μέλη του IEA, ε, παρόλο που δεν είναι μέλη του NPT. Ε, Οι αποφάσεις κυρώσεων λοιπόν παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και εκεί τα πράγματα αλλάζουν διαφορετικά. Και βεβαίω η παγκοσμιοποίηση έχει και αυτή κατά πάσα πιθανότητα διαδραματίσει το ρόλο τη, διότι πολλοί όσοι παρέχουν αυτήν την πυρηνική τεχνολογία τη σήμερα ημέρα να έχουν διαφορετικά πολιτικά, οικονομικά κίνητρα και συμφέροντα. Οπότε η κατάσταση είναι διαφορετική από ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Για τις μελλοντικές προοπτικές της NPT. Τι μπορούμε να πούμε. Ερώτημα κλειδί και το ανέφερα προηγουμένως για τα χημικά και βιολογικά όπλα. Το ερώτημα κλειδί είναι λοιπόν η NPT μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον όπου τα πυρηνικά όπλα έχουν κάποια έστω και περιθωριακή ή περιφερειακή νομιμότητα ως αποτρεπτικά. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ωφελούνται τις συνεργασίες στον πυρηνικό τομέα και έχουν πυρηνικά όπλα αλλά δεν συμμετέχουν στην NPT. Και το ΔΕΚ, μάλλον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του 1996 που στη συμβουλευτική της απόφαση άφησε μισάνοιχτη την πόρτα λέγοντας ότι τα πυρηνικά όπλα μπορεί να θεωρούνται και νόμιμα σε ορισμένες περιπτώσεις όταν διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση ενός κράτους ή έθνους. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να στραφούμε στο άρθρο 6 της NPT, αφοπλισμός. Είναι βασικό ζήτημα αυτό που μπορεί να αποτελέσει κλίδα της επιτυχίας του χρόνου στην διάσκεψη για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της κατάστασης Πάντως το καθεστώς ε, παρακολούθησης και ελέγχου του οπλισμού είναι κατακαιρματισμένο. Υπάρχουν διάφορα στάδια του, της διαδικασίας οπλισμού που διέπονται από διαφορετικές συνθήκες διεθνείς ή περιφερειακές, ορισμένα θέματα εφαρμόζονται, άλλα έχουν παγώσει γιατί αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης επί χρόνια, ξεκινούν και διακόπτονται διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής. Ένα ενδεχομένως απλό βήμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ένα πρώτο βήμα για την επιβίωση της NPT στο μέλλον είναι η προσπάθεια διαπραγμάτευσης για απαγόρευση χρήσεως των πυρηνικών όπλων. Χρήσεως, όχι κατοχής και απόκτησης, αλλά χρήσης, με βάση το πρωτόκολλο της Γενέβης του 1925. Μονοσέλιδο κείμενο δεν μιλάει, δεν είναι συνθήκη αφοπλισμού. Έχει παραβιαστεί βεβαίως μία-δυο φορέ για τα χημικά όπλα, αλλά συγχρόνω ε, κατέστησε πολύ δύσκολο για αυτούς που θέλουν να προωθήσουν τα χημικά και βιολογικά όπλα να δικαιολογήσουν στην, στο στρατιωτικό σκέλος ότι είναι νόμιμο μέσο άμυνας. Μας πήρε χρόνο, άρα μπορέσαμε να το αποκλείσουμε. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, μια απαγόρευση τη χρήση των πυρηνικών όπλων επί τη βάση του πρωτοκόλου θα μπορούσε να είναι μια λύση. Με όχι επαχθή δηλαδή διαδικασία διαπραγματεύσεων και όλα τα κράτη θα πρέπει να την προσυπογράψουν από την αρχή. Το πρωτοκόλλο της Γενέβη μπήκε το 1928, αλλά τα Ηνωμένε Πολιτείε ε, μόνο το 1975 ε, ε, το ασπάστηκαν, προσεχώρησαν για να το πω έτσι. Αυτά. Ας βάλω μια τελεία εδώ και να σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σας. Εγώ σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Δίδω το λόγο στον κύριο Μάιερ. Um, ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με καλέσατε να μιλήσω σε αυτή την ακρόαση και είναι πολύ καλή η ε, συγκυρία της συναντήσεως αυτής εφόσον πρόκειται να συζητήσουμε ε, την ε, εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας άρα αυτό είναι πολύ βασικό για το θέμα της συνθήκης για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων την NPT και τη διασύνδεσή της με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, τα τελευταία χρόνια άλλωστε έχει, ε, ε, έχει επιβεβαιωθεί ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να συμβάλλει σε μια επιτυχή συνάντηση διότι στο ψήφισμα 80-87 έχει υιοθετηθεί η μη διάδοση πυρνικών και ε, τώρα είναι συντονισμένες οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κοινό πρόγραμμα για τη μη διάδοση πυρνικών όπλων και σχάσιμων υλικών. Του χρόνου μάλιστα θα υπάρχει αναθεωριστική διάσκεψη ε, και η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει νέες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική στο θέμα της μη διάδοσης. Επιπλέον υπάρχουν ορισμένες ε, προκλήσεις οι οποία πρέπει να ενισχύσει ε, την προβολή της και όπως ε, ήδη είπε ο προηγούμενος ομιλής σας, Υπάρχουν πολλές χώρες με πυρηνικά όπλα που δεν έχουν υιοθετήσει ε, τον στόχο της καταργήσεως των πυρηνικών όπλων. Τα θέματα με το Ιράν και την Κορία δεν έχουν λυθεί και ε, το, Ιράν ε, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα διότι Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια διαλόγου. Υπάρχουν άλλωστε και άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή που χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ενεργείας και ε, μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και ε, να υπάρξει μια κακή χρήση και αρνητική χρήση των πυρηνικών ε, δυνατοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ στις διάφορες λειτουργίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία στο παρελθόν έχει ηγηθεί ε, ως παράδειγμα και ως πρότυπο και ε, έχει ε, αποτελέσει έναν προπομπό για συμφωνίες καταργήσεως των πυρνικών οπλισμών και έχει προσπαθήσει να συγκεράσει απόψεις αντιμαχόμενες και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το νέο πολιτικό ο πλαίσιο το οποίο επηρεάζει την κατάσταση της NPT, του σχετικού συνεδρίου και πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει την έκβαση του χρόνου. Υπάρχει ένα γραπτό κείμενο ε, των παρατηρήσεών μου το οποίο θα σας δώσω στη συνέχεια της συνεδριάσεως όπου θα δείτε ότι αναφέρομαι πιο λεπτομερώς σε διάφορα θέματα. Ε, υπάρχει ένα πρότυπο και πρέπει εδώ να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μία εξαιρετική θέση και υπάρχουν διάφορες δυνατότητες οι οποίες ε, επιτρέπουν ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθηθεί ε, και γενικώς πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπόρεσε να ε, τοποθετηθεί σχετικά με ε, τις σχέσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ινδίας επί του θέματος και ήταν μια βασική αποτυχία για τη στρατηγική μη διαδόσεως των πυρνικών όπλων και μέχρι του χρόνου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ε, θα ε, υπάρξουν ε, και άλλες επιπτώσεις και επιπλέον η υπάρχει θέμα ε, μεταδόσεως της πυρηνικής τεχνολογίας προς τρίτες χώρες, προς τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση προς την Αφρική παραδείγματο χάρη. Ε, υπάρχουν ορισμένες τεχνολογίες οι οποίες είναι ευαίσθητες όπως ο εμπλουτισμός του ουρανίου και του πλουτονίου και ε, υπάρχει μία προσπάθεια περιορισμού της γενικότερης διάδοσης αυτών των μεθόδων μέσω των συμφωνιών ε, για τη μη διάδοση των ε, πυρηνικών ε, δοκιμών. Πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε αυτές τις δυνατότητες πυρηνικών οπλισμών με τους συμβατικούς και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Καταρχήν όσον αφορά την ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να έχουμε μία πιο αποτελεσματική πολιτική και να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας με πιο αποτελεσματική αμυντική συνεργασία όσον αφορά τον έλεγχο των οπλισμών διότι ε, αναφερόμαστε στην άμυνα στο κείμενο 54 φορές χωρίς όμως να αναφερόμαστε στην, στον αφοπλισμό ή στη συνεργασία. Πρέπει λοιπόν οι κινήσεις αυτές να αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο του, της εντολής του νέου υπάτου εκπροσώπου τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποτελέσει το επίκεντρο όλων των προσπαθειών για την ε, ανάσχεση της, ε, επεκτα... της διαδόσεως των πυρηνικών ε, οπλισμών στο παρελθόν έχουμε δει ότι ε, το καθεστώς ε, ε, μπόρεσε να βοηθήσει όταν, όταν κατά τη διάρκεια της κυβερνήσεως Μπούς, δηλαδή κατά την τελευταία οκταετία. Γενικότερο όμως η πολιτική αυτή έχει αλλάξει πάρα πολύ ε, λόγω της αλλαγής πολιτικής της Washington και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προσπαθήσει να ενισχύσει τις διεθνείς οργανώσεις μη διαδόσεως μέσω χρηματοδοτήσεως και εδώ επανέρχομαστε εις ε, τις προειδοποιήσεις του Μοχάμετ Ελμπαραντέη ε, ε, ο οποίος είχε ζητήσει να διπλασιαστεί χρηματοδότηση κατά την επόμενη τετραετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να υιοθετήσει αυτή την πρόταση και άλλωστε ορισμένες χώρες ε, συμφωνούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας ενώ ίσως θα χρειαστεί να ενισχυθούν περισσότερο. Όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια για να προλάβουμε ε, την πυρηνική τρομοκρατία που είναι ένας πολύ βασικός τομέας. Ε, πρόκειται 12 και 13 Απριλίου να γίνει μια σχετική διάσκεψη στη Washington για να διατυπωθούν νέα μέτρα καλύτερης συνεργασίας και θα έπρεπε να βοηθήσουμε τους στόχους ε, του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος ε, θέλει να ενισχύσει τις σχετικές προσπάθειες την επόμενη τετραετία. Άλλωστε, ε, θα πρέπει στα πλαίσια της NPT να αποτελέσει η προσπάθεια αυτή τον τέταρτο πυλώνα και ε, ε, να ε, υπάρξει μία συζήτηση για τους τρεις άλλους πυλώνες. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποια μεσολάβηση και έχει παίξει ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση διότι ε, στις ε, διάφορες ε, συζητήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να ακολουθήσει μία μέση οδό και να ενισχύσει την συνθήκη. Από τη μία πλευρά υπήρχαν όμως, υπήρχε η κυβέρνηση Μπούς και από την άλλη πλευρά ορισμένες ε, ε, μη ενταγμένες ε, χώρες και χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος της NPT ενώ υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσει, να εμποδίσει τη συμφωνία αντί να την προωθήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, ενισχύσει τον ε, ρόλο της ε, σαν διαμεσολαβητής ενισχύοντας τις αποφάσεις του 2005 για τον έλεγχο των οπλισμών και αναγνωρίζοντας το δεσμευτικό χαρακτήρα των ήδη συμπεφωνημένων εγγράφων κατά τη διάσκεψη του 2002 Οπότε υπήρξε το πρόβλημα για τη Γαλλία η οποία είχε αμφισβητήσει τις προηγούμενες συμφωνίες επί του θέματος σχετικά με ε, τα σχάσιμα υλικά. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να κοιτάξουμε ε, ποιες άλλες δυνατότητες υπάρχουν για προώθηση των στόχων μας και υπάρχει και ένα διαδικαστικό θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει κανείς ε, να επιτύχει και ε, ή στο παρελθόν έπρεπε να υπάρξει συμφωνία όλων των κρατών μελών ενώ τώρα εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πιο θετική διότι ο πρόεδρος Πρόεδρος και ε, ο ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν να έχουν έναν πιο επικοδομητικό ε, ρόλο και ε, θα έπρεπε να τους δοθεί μια πιο ευρεία εντολή ώστε κατά την αναθεωρητική διάσκεψη να μπορέσουν να συμβάλλουν. Ε, για να μπορέσει να υπάρξει υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών μέτρων και πιο αυστηρών ε, προδιαγραφών για την πυρηνική τεχνολογία. Θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ε, τον, τον επικεφαλής της προσπαθίας αυτής. Ε, πρέπει να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση Ομπάμα έχει συμβάλει ριζικά σε μία βελτίωση, αλλά μέχρι στιγμής ε, η στρατηγική που είχε διατυπωθεί η στο δεύτερο ήμιση του 2008 υπό Γαλλική Προεδρία είχαν οδηγήσει σε μια περιορισμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΕΠΑ και είπα επί ενός κειμένου που συμφωνήθηκε για περιορισμένα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως εντωμεταξύ ακόμη ε, δεν ε, έχει απαντήσει στην πρόσκληση του Προέδρου Ομπάμα για περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Μέχρι στιγμής δεν έχω αναφερθεί στη γενική θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον αφοπλισμό και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι κινήσεις μπορεί να θεωρηθούν ε, ανεπαρκείς εάν η Ευρώπη θέλει να συμβάλλει Πρέπει να αναφερθεί σε συγκεκριμένα θέματα στο εάν δηλαδή η κατάργηση των πυρηνικών οπλισμών είναι εφικτή και επιθυμητή, αν μπορεί να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και να καταρτήσει μία ημερήσια διάταξη η οποία θα αποτελέσει τη βάση ε, μίας συζητήσεως μεταξύ των ε, κρατών για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Εφόσον όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τούδε ποτέ με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να ξεκινήσει επί μηδενικής βάσεως και έτσι ε, μπορεί να υπάρξουν διαβουλεύσεις ε, σε διάφορες ομάδες εργασίας ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Κοινωνίας των Πολιτών. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συζήτηση των πυρηνικών θεμάτων. Για να συνοψίσω τώρα. <clears throat> Εδώ και πάνω από μισό χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει μια μοναδική δυνατότητα της Ένωσης να ενδυναμώσει, να προωθήσει την εφαρμογή του καθεστώτος μη διάδοσης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να τα προβλάβουμε όλα αυτά βέβαια για την αναθεώρηση του Μαΐου. Ευχαριστούμε κύριε Μέγερ για την παρουσίαση αυτή των στόχων της Μίδας ΤΕΝΠ συνθήκης μη διάδοσης, και γιατί τα συνδέσατε λίγο με την τωρινή πολιτική κρίση σε σχέση με το Ιράν ιδίως. Ο επόμενος. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Πιστεύω και εγώ ότι αυτή η δημόσια ακρόαση είναι κάτι το ιδιαίτερα ε, σωστό για, όχι μόνο εν ώψη της αναθεώρησης της συνθήκης μη αλλά και λόγω των κρίσεων με το Ιράν και την Κορέα. Θα βασιστώ σε μια παρουσίαση της κατάστασης στο Ιράν και στη Βόρεια Κορέα, αλλά επίσης θα μιλήσω για τις επιπτώσεις του καθεστώτος μη διάδοσης <clears throat> γενικότερα. Γιατί η διάσκεψη του 2010 δεν, πρέπει να, δεν μπορεί να αγνοήσει τις δύο αυτές κρίσεις αν δεν θέλει να υπάρξει σημαντική λάθος και διστρέβλωση των στόχων της συνθήκης. Λοιπόν, ένα γενικότερο ιστορικό για την κρίση με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Καταρχήν, ως προς την ορατότητά τους, για να το πω έτσι, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι παλιό και γνωστό πρόβλημα. Οι βορειοκορεατικές και ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ήδη από τη δεκαετία του 70 είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται με διαφορετικούς ρυθμούς. Υπήρξαν επιταχύνσεις τη δεκαετία του 90 και ε, έφτασαν σε φάση ανοιχτή κρίσης μετά το 2000. Δεν είναι λοιπόν τίποτε μείζονες ε, κρίσεις αλλά παλαιές και γνωστές αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεύτερον, για την ίδια τη διπλωματική κρίση μέσα στη λογική αυτή της μακράς διαρκείας, το να προσπαθήσουμε να πείσουμε τη Βόρεια Κορέα, οι προσπάθειες να πιστεί η Βόρεια Κορέα να μην κάνει τέτοια πειράματα είναι και αυτές παλιές. Το 2003 είχε δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από τη συνθήκη αλλά μετά οι Ηνωμένε Πολιτείε ιδιαίτερα προσπάθησαν να κάνουν διαπραγματεύσει για να πείσουν τη Βόρεια Κορέα να αλλάξει γνώμη. Από το 2003 άρχισε να εφαρμόζεται μια διαδικασία συνεννόηση έξι κρατών με την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες βέβαια και την Κορέα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα αλλά δεν πέτυχε τίποτα η προσπάθεια αυτή μέχρι τώρα. Για το Ιράν η κρίση θεωρείται έκδηλη από το 2003, από τότε δηλαδή που φάνηκε ότι το Ιράν έχει κρύψει εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, δεν τις έχει δηλώσει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας. Από το 2003 λοιπόν βλέπουμε ότι η κρίση αυτή συνεχίζεται γιατί ανακαλύπτονται και άλλες αδήλωτες εγκαταστάσεις και υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας. Αυτή λοιπόν η κρίση ε, είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τις συνήθεις διπλωματικές κρίσεις. Οι δύο κρίσεις αυτές, Κορέα και Ιράν, είναι ανησυχητικές διότι δείχνουν ότι υπάρχουν νέα φαινόμενα που τα είχαμε υποτιμήσει στην συνθήκη μη διάδοσης προηγουμένως. Πρώτον, υπάρχει μια διάδοση νότου-νότου. Στην περίπτωση του Ιράν, το Ιράν έλαβε τεχνολογίες διάδοσης από το Πακιστάν μέσω του δικτύου EQCAN. Και στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας, που είναι ο κύριος πολιτής βλημάτων στο Ιράν και άλλες χώρες, ε, μόνη της τα έκανε όλα. Είναι λοιπόν θέμα νότου-νότου. Και αλλάζει ριζικά την κατάσταση που ίσχυε τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή το καθεστώς ελεγχομένων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνολογιών. Προηγουμένως η διάδοση συνήθως γινόταν από εγκαταστάσεις των βιομηχανικών χωρών, ενώ σε αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχει μεταφορά τεχνολογίας νότου-νότου. Δεν μπορούν δηλαδή πλέον οι βιομηχανικές χώρες Δυτικές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς, Ηνωμένε Πολιτείες ή ακόμη και η Ρωσία να ελέγξουν τη μεταφορά αυτή τεχνολογίας. Δεύτερον, επίσης πολύ ενισχυτικό, η διάδοση αυτή γίνεται από κράτη που έχουν συνυπογράψει τη συνθήκη μη διάδοσης και τα δύο και που άρα την παραβιάζουν και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό διότι πάλι πριν από 30 χρόνια, εδώ και 30 χρόνια μάλλον, στόχος ήταν πώς θα διασφαλίσουμε οι περισσότερες όσο δυνατόν χώρες να υπογράψουν τη συνθήκη. Τώρα όμως έχουμε χώρες όπου έχουν υπογράψει τη συνθήκη ήδη, αλλά δεν την εφαρμόζουν και αναπτύσσουν στρατιωτικού χαρακτήρα προγράμματα παρά την υπογραφή τους. Άρα δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους, αλλά επίσης αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο που μπορεί να διαβρώσει και άλλες χώρες. Ξεπερνάει κατά πολύ το καθαρά πυρηνικό θέμα, μπορεί να αφορά και τη συνθήκη για τα βιολογικά ή χημικά όπιλα. Οι μηχανισμοί ελέγχου για τα πυρηνικά θεωρούνται πιο βέβαιοι και σταθεροί και σίγουροι από ότι στις άλλες περιπτώσεις, αν και αυτό δεν είναι σίγουρο γιατί δεν έχουν γίνει έλεγχοι για τα χημικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Υπάρχουν και άλλα προηγούμενα και στη δεκαετία του 80 είχε προσπαθήσει το Ιράκ να διαπράξει διάδοση και η Λιβύη μέχρι το 2000 και υπήρξαν και ορισμένες ανησυχίες για προγράμματα της Συρίας πάντα από χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Τέταρτο στοιχείο. Εδώ βλέπουμε, διαπιστώνουμε μια παραβίαση της συνθήκης μη διάδοσης και των εγγυητικών συμφωνιών. Διπλή παραβίαση, γιατί υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες ή μη δεδηλωμένες που αποτελούν άρα παραβίαση των υποχρεώσεων των υπογραφών της συνθήκη, επίσης παραβίαση των κανόνων απόσυρσης Και αυτό το λέω διότι νομίζω ότι η απόσταση της Βόρειας Κορέας δεν έγινε νομοτύπος, δεν σεβάστηκε το άρθρο 10. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πλέον ότι η Κορέα είναι χώρα που σέβεται τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, γιατί ο πρόεδρος προηγουμένως είχε πει ότι, ο κύριος Αντέρς μάλλον προηγούμενος ομιλητής είχε πει ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Κορέα για την προετοιμασία της διάσκεψης του 2010. Οι παραβιάσεις αυτές για το, Ιρά, για το Ιράν, για τον εμπλουτισμό του ουρανίου, οδήγησαν σε διαμαρτυρίες της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενεργείας και του Συμβουλίου Ασφαλείας γιατί υπήρξε διαπίστωση πολλαπλών παραβιάσεων. Αυτές οι κρίσεις είναι επίσης ανησυχητικές ως προς το θέμα της διάδοσης τεχνολογιών. Περισσότερο στην Κορέα και λιγότερο στο Ιράν βλέπουμε ότι οι χώρες δεν διαδίδουν απλώς πυρηνικές εγκαταστάσεις αλλά μπορούν την τεχνολογία που αναπτύσσουν να τη χορηγήσουν και σε άλλες τρίτες χώρες. Αυτό το κάνει η Κορέα για τα βλήματα, αλλά υπάρχουν ανησυχίες και για τα πυρηνικά, όπως κάνει και το Πακιστάν, το οποίο όμως δεν έχει συνυπογράψει. Προσθέτω ότι οι ανησυχίες και οι απειλές αυτές δεν είναι μόνο τοπικές αλλά σφαιρικές, καθολικές. Δηλαδή, δεν θα ήταν σωστό οι Ευρωπαίοι να θεωρήσουν ότι η Ιρανική ή η Βορειοκορεατική βόμβα είναι απειλή μόνο για τις γειτονικές της, τους χώρες. Μπορούν να απειλήσουν και χώρες πολύ μακρύτερα. Και έχει γι' αυτό επιπτώσεις και για τη δική μας ασφάλεια και την ασφάλεια δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, τελευταίο, πώς να διαχειριστούμε τις κρίσεις αυτές. Εδώ έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση στα όρια της διπλωματίας. Όλοι είμαστε υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, αλλά βλέπουμε και στη διαδικασία των λεγόμενων six party talks και στη διαδικασία για την Κορέα και στη διαδικασία ε3 συν 3 ή συν 1 κτλ ανάλογα με το πώς το ονομάζει κάθε πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για συνεννόηση με τις χώρες αυτές ως προς τα πυρηνικά καθυστερούν και δεν έχουν μέχρι τώρα αποφέρει τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα διότι μια αποτυχία της διπλωματίας θα σήμαινε ότι όσοι έχουν τον πειρασμό να εφαρμόσουν στρατιωτικές λύσεις ε, ε, έχουν ακόμη περισσότερο, βαρύνει περισσότερο η γνώμη τους. Και αυτό βλέπετε ότι μπορεί να αποτελέσει χειροτέρευση των κρίσεων. Μετά το τέλος το δεύτερο. Οι κρίσεις αυτές είναι άμεση απειλή για το μέλλον της συνθήκης μη διάδοσης. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μερικές χώρες να θεωρήσουν ότι η σημίδα, η συνθήκη μη διάδοσης και η Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ασφαλείας, τα δύο θεμέλια δηλαδή για την ποινική ασφάλεια διεθνώς, είναι αποτυχία. Μετά από 40 ετή, 40 ετή επιτυχία αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε στην προετοιμασία της διάσκεψης του 2010, αν και δεν θα συζητήσει αποκλειστικά τις κρίσεις αυτές, ούτε έχει στόχο να τις λύσει. Αλλά πάντως είναι σημαντικό να λάβει υπόψη της τα θέματα αυτά της κρίσης δηλαδή. Μετά το δεύτερο λοιπόν, το δεύτερο δεύτερο. Η συνθήκη μη διάδοσης μπορεί να αφορά και τα πυρηνικά και τα χημικά και τα βιολογικά όπλα. Αν δηλαδή δεν μπορέσουμε να διαπιστώσουμε με αποδείξεις τις παραβιάσεις και δεν μπορέσουμε και να απαντήσουμε σε αυτές με το δια της διπλωματικής οδού, τότε μπορεί μερικές χώρες που θεωρούν ότι η συνθήκη μη διάνοησης είναι και εργαλείο για συλλογική ασφάλεια που πρέπει να χορηγεί ορισμένες εγγυήσεις ότι οι γείτονέ τους δεν διαδίδουν, τότε μπορεί οι χώρες αυτές να βγάλουν αρνητικά συμπεράσματα για την ίδια τη συνθήκη. Και μπορεί δηλαδή προοδευτικά ή απότομα να μην υπάρχει πλέον καμία αξιοπιστία της συνθήκης και να καταστραφεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αν υπάρξει και δεύτερη απόσυρση όπως της Βορείας Κορέας. Αν το Ιράν καταφέρει να πετύχει τους στρατιωτικούς του στόχους χωρίς να φύγει από τη συνθήκη, ε, θα έχει ήδη αποδυναμώσει τη συνθήκη. Η προοδευτική καταστροφή της συνθήκης τώρα θα ήταν προοδευτική μείωση της αξιοπιστίας της και της εμπιστοσύνης των συμβαλωμένων μερών. Και τελικά η καταστροφή της συνένεσης 289 ετών για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Έπειτα πέρα από το ίδιο το καθεστώς η κρίση αυτή θέτει το πρόβλημα μιας αλυσιδωτής ε, διάδοσης δηλαδή μιας νέας, ενός νέου αγώνα δρόμου για τους εξοπλισμούς. Ορισμένες χώρες στη Μέση Ανατολή και στην Άπο Ανατολή, όπως και στην Νοτιοανατολική Ασία, αναρωτιούνται για τα, το μέλλον των πυρηνικών ή εξοπλιστικών των προγραμμάτων αν δεν έχουν την εγγύηση ότι οι μεγάλοι ή μικροί γειτονέ του ε, δεν διαδίδουν πυρηνικά όπλα, τότε μπορεί να αναρωτηθούν μήπως πρέπει να βρουν κάποια άλλη καλύτερη λύση για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους ή να συνάψουν συμμαχίες και συμφωνίες με πυρηνικές δυνάμεις ή απλώς να σκεφτούν την εφαρμογή ενός δικού τους εθνικού πυρηνικού προγράμματος για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή των γειτόνων τους. Στην Τουρκία, στην Ιαπωνία γίνονται δημόσιες συζητήσεις για τα θέματα αυτά και αυτά που λέγονται είναι ανησυχητικά. Υπάρχει επίσης ένας πραγματικός κίνδυνος χρήσης, πραγματικής χρήσης του πυρηνικού όπλου. Διότι αν συνεχιστεί η διάδοση τότε αυξάνεται ο κίνδυνος πραγματικής χρήσης του πυρηνικού όπλου είτε από τρομοκράτας είτε από κράτη. Ίσως και ως απάντηση σε απειλές από κράτη-μέλη της συνθήκης μη διάδοσης, αν πάψει να υπάρχει το πυρηνικό ταμπού. Το τελευταίο σημείο το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο των επομένων συζητήσεων ε, σε έναν ε, κόσμο με, απο... με επιτυχημένη <clears throat> συμφωνία μη διαδόσεω πυρηνικών όπλων δεν θα υπήρχαν νέες πυρηνικές δυνάμεις των οποίων η παρουσία αποδυναμώνει την προπτική της ε, επιδιώξεως δημιουργίας ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Οπότε για να προσπαθήσω να καταλήξω τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ίσως είναι ε, η κατάλληλη στιγμή να πάρουμε πολύ στα σοβαρά τις δύο αυτές κρίσεις. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν διπλωματίες και χώρες που ασχολούνται ενεργά με τα θέματα αυτά και δεν τις αμφισβητούμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές χώρες, ιδίως εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θεωρούν ότι η υπόθεση του Ιράν ε, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται για να δούμε εάν το Ιράν μπορεί να έχει ε, πυρηνική τεχνολογία και πρόκειται για μια ε, κεντρική δικτατορία η οποία αναλαμβάνει υπερβολικές ενέργειες ενώ θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά τις κρίσεις αυτές σε όλα τα κράτη του ο κόσμου και γι' αυτό ίσως η επόμενη διάσκεψη θα μας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό και να πείσουμε ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να υπογράψουν τη συμφωνία TNP, χώρες δηλαδή ε, σαν ε, την Βραζιλία και άλλες για να κινητοποιηθούν και να τους ε, τονίσουμε ότι αυτά τα θέματα μας απασχολούν ιδιαίτερος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία στο TMP. Υπάρχουν ε, τρεις ε, ε, πτυχές εις τη συμφωνία αυτή και πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα μέτρα τα οποία υπάρχουν κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία συμφωνία ε, με μόνο έναν, με μία εξαίρεση που θα είναι ενδεχομένως το Ιράν εάν δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέλος της συμφωνίας αυτής. Εάν όμως καταστούν υποχρεωτικές ε, οι επιπρόσθετες πράξεις ε, και συμφωνίες του Οργανισμού Πυρηνικής Ενεργείας ε, θα μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε καλύτερα και η πρώτη κίνηση του Ιράν ήταν να εγκαταλείψει την εφαρμογή των επιπροσθέτων πρωτοκόλων. Πρέπει να αποφύγουμε την απόσυρση από το TNP και δεν βλέπουμε γιατί θα έπρεπε έπρεπε μία χώρα να μπορεί να απόσχει όπως το έκανε η Βόρειος Κορέα και να μπορεί συγχρόνως να υποφελείται από 20 χρόνια πυρηνική συνεργασίας όπως έγινε με το Ιράν και μετά από 20 χρόνια μας πει τώρα άλλαξα γνώμη και τώρα θα αναλάβω ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα και το μόνο που χρειάζομαι είναι να αποσυρθώ από τη συμφωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάσκεψη του 2010 για να υπάρχει μία ενισχυμένη προσπάθεια μη επεκτάσεως ε, και για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες τις ε, παράνομες διακινήσεις ε, πυρηνικών όπλων μία μη επέκταση η οποία θα είναι ισχυρή και θα προσφέρει εχέγγυα σε διάφορες χώρες ε, θα επιτρέψει στις νότιες χώρες να μπορέσουν ε, να δεχθούν μεταφορά τεχνολογίας χωρίς όμως να αποβλέπουν στη διάδοση και να δούμε ε, τα κράτη τα οποία έχουν ήδη πυρηνικά όπλα να μπορέσουν να εφαρμόσουν το άρθρο 6 για τον αφοπλισμό κατά τρόπον ώστε τα κράτη αυτά να μπορέσουν να προχωρήσουν και καταλήγω με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα έλεγα ότι σχετικά με την Βόρειο Κορέα ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι περιορισμένος όπως ίσως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει πρέπει να ε, χρειάστηκε ε, να ε, να πληρώσει για την προηγούμενη συμφωνία, πράγμα το οποίο τώρα απορρίπτει. Παραδείγματο χάρη δεν θα στηρίξει το καθεστώς Βορείας Κορέας χωρίς αντικρίσματα και θα πρέπει ε, με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει και τη Βόρειο Κορέα ή στην επόμενη συμφωνία. Θα πρέπει άλλωστε και η Κίνα και η Ρωσία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες να συμμετάσχουν για να υπάρχει μια κοινή προσπάθεια, να μην είναι ένας από φάκελος τον οποίο επιζητούν και να μπορέσει να αποδείξει την ανησυχία της για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Για το Ιράν ο ρόλος είναι πολύ πιο γενικός διότι υπάρχουν τρεις, προ... τρεις χώρες ε, οι οποίες προσπαθούν ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ε, βασικό θέμα και ε, το Ιράν θα πρέπει ε, να αποτελέσει έναν ε, σοβαρό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για τη Βόρειο Κορέα. Θα πρέπει λοιπόν να μην αποκλείσουμε τις ε, δυνατότητες των κυρώσεων ε, ευρωπαϊκών εάν ε, τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να υιοθετήσουν ένα πιο σαφές σύστημα κυρώσεων όταν ο κύριος Αχμαντινετζάν μας ζητά να ε, μας, λέει, μας ανακοινώνει ότι αυξάνει τις προσπάθειες εμπλουτισμού ε, πέραν των εγκαταστάσεων τις οποίες ανακαλύψαμε ε, προσφάτως και δεν θα πρέπει να δεχθούμε τέτοιες κινήσεις. Και τελειώνοντας, συμφωνώ με τον κύριο Μάγερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξει και έχει ένα του για να... και εφόσον εγώ ο ίδιος έχω έχω συμμετάχει με τη γαλλική αντιπροσωπεία σε διάφορα συνέδρια. Ξέρω ότι όταν μπορεί να καταργεί... Να, προχωρήσει η η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με ολόκληρη την οικογένεια του TNP θα πρέπει να έχει μία φιλόδοξη πολιτική και στόχη τους οποίους θα επιζητήσει μέσω αυτής της ε, διασκέψεως και για τον αφοπλισμό και για ε, την ε, ειρηνική προώθηση των ποινικών δυνατοτήτων και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην κυρία Ρεμπέκα Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόνζο και την Υποπιτροπή για την ασφάλεια και την άμυνα για μια πολύ κέρια, πιστεύω, ακρόαση που θα ακολουθηθεί και από άλλες. Και βεβαίως σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Νομίζω ότι άπαντες οι παριστάμενοι έχουν επίγνωση του ότι τον Απρίλιο του 2009 ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε μια πολύ σημαντική ομιλία στην Πράγα για τα όπλα, στην οποία ανέφερε και κατά λέξη παραθέτω σαφώς και με πεποίθηση η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εξεύρει ρήνη ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς πυρηνικά όπλα. Τέλος της παράθεσης. Έτσι μετακινείται από μια σειρά δεκαετιών πολιτικής επιζήτησης πυρηνικών και διαχείρισης του πυρηνικού πλαστασίου προς μια κατεύθυνση κατάργησης αυτών. Όπως ανεγνώρισε ο Ομπάμα σε μια άνευ προηγουμένου συνάντηση του Συμβουλίου της Ασφαλείας ε, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2009 που οδήγησε στην ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ψηφίματος 1887 υπήρχε, υπήρχαν οι τέσσερις ε, υπότες οι λεγόμενοι οι οποίοι έγραψαν στην Wall Street Journal τον Ιανουάριο του 2007 ότι η εξάρτηση ε, στα, από τα πυρηνικά γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη και όλο και λιγότερο αποτελεσματική ως αποτρεπτικό, ως μέσο αποτροπής του πολέμου. Η στροφή αυτή λοιπόν μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι σαφώς πιο ρεαλιστική από την αφελή και ομφαλοσκοπική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η διάδοση των πυρηνικών όπλων μπορεί να συνεχιστεί αενάως χωρίς να παραδεχτούμε όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα ότι η χρήση των πυρηνικών όπλων είναι αναπόφευκτη. Με την έκκληση του για πυρηνικό αφοπλισμό ο πρόεδρος Ομπάμα υπενθύμησε ότι αν εκραγεί μία πυρηνική βόμβα στη μία άκρη του κόσμου, θα μπορούσαν στην άλλη άκρη του κόσμου να σκοτωθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Όπου και αν γίνει δεν υπάρχει τέλος των τραγικών συνεπειών για την συνολική ασφάλεια, για την κοινωνία, την οικονομία και βεβαίως εσχάτως την επιβίωσή μας. Και αυτό που ήταν παράθεση, θα πρέπει να το επαναλάβουμε, διότι με τον ψυχρό πόλεμο και ε, στην Ευρώπη ιδιαίτερα ε, είμαστε εφησυχασμένοι. Αυτάρισκα σχεδόν αποδεχόμαστε την ύπαρξη των πυρηνικών όπλων. Το ερώτημα λοιπόν το το θέμα το οποίο θέτω είναι ότι υπάρχει ρεαλιστική πεποίθηση για το ότι αυτό το status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για πρώτη φορά το γνώρισε ο πρόεδρος Ομπάμα και συμφωνώ μαζί του. Το status quo δεν είναι ισορροπημένο. Ενέχει, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ότι θα χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Ότι μια πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίπεινα και άρα σε κλιμάκωση. Και ενέχει τον κίνδυνο αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλά πυρηνικά όπλα σε έναν περιφερειακό ή συνολικό παγκόσμιο πόλεμο οι νεκροί δεν θα μετρούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Όπως λοιπόν ανησυχούμε για την κλιματική μεταβολή, θα πρέπει να ανησυχούμε της ακτινοβολίας από διάφορες, όχι μία, από διάφορες πυρηνικές ε, εκρήξεις που δεν είναι ανάγκη να είναι και πολλές όπως λένε οι επιστήμονες ειθύνοντες περί το περιβάλλον. Μαζική πείνα, θα προκαλέσει εκτός από τους θανάτους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από το υφιστάμενο ήδη πυρηνικό οπλοστάσιο, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να αυξηθεί, η να διαδοθεί περισσότερο. Άρα, άρα, ερωτώ, η ασφάλεια σε έναν κόσμο πυρηνικών όπλων είναι ρεαλιστική. Η απάντηση βεβαίως είναι αρνητική. Έχω αφιερώσει μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου υπέρ του αφοπλισμού γιατί πιστεύω ότι τα πολύνικα όπλα είναι ανήθικα, αναξιόπιστα και σαθρά θεμέλια για την αποτροπή του πολέμου. Επί τη βάση κάποιων αφελών και α, τσαρλατάνικων πεπιθήσεων οι οποίες μόνο κακό μπορούν να προκαλέσουν στο εγγύς μέλλον που μπορεί να είναι καταστροφικό με την χρήση των πυρηνικών όπλων. Και θεωρώ ενδιαφέρον το γεγονό ότι αν όχι και οι τρει, τουλάχιστον δύο από του προλαλήσαντε έθεσαν το συγκεκριμένο ερώτημα. Για τη χρήση δηλαδή των πυρηνικών όπλων. Ω εκ τούτου είναι ανακούφιση που ακούμε τον ε, ε, Μπάρακ Ομπάμα, τον Γκόρντον Μπράουν και άλλου ηγέτε ε, του κόσμου να ομιλούν πλέον για αφοπλισμό ως αποτροπή. Και συμπεριλαμβάνω και τον Χένρι Κίτσιντζερ και τον κύριο Γκορμπατσόφ. Διότι η συνεχιζόμενη κατοχή και διάδοση πυρηνικών όπλων οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας. Εμείς θέλουμε ένα κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά. Η, η πρώτη δοκιμή για το αν το εννοεί αυτό που λέει ο πρόεδρος Ομπάμα είναι η αναθεώρηση, η αξιολόγηση της ε, αμερικανο-ρωσικής σχέσεως. Όχι μόνο το Start Plus που ελπίζουμε ότι θα ε, υπογραφεί πριν εκπνεύσει το προηγούμενο, αλλά τι θα το ακολουθήσει. Είναι σαφές ότι οι ηγέτες στον κόσμο θα πρέπει να κάνουν βεβαίως πολλά περισσότερα για να περάσουν αυτό το μήνυμα. Το όραμά τους θα πρέπει να το μετατρέψουν σε πρακτικές προτάσεις. Ουδόλως εύκολο. Αλλά το σύστημα αυτό που έχει κυριαρχήσει τώρα και που έχει επικρατήσει και το οποίο θεωρείται ε, ότι προωθεί ένα καθεστώς μη διάδοσης, οδηγεί πολύ συχνά στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ένα μικρός αριθμός κρατών θεωρεί τα πυρηνικά όπλα ως μια, ένα τεράστιο ατού, ενώ ο υπόλοιπο κόσμος τα έχει αποκλείσει. Προκύπτει αυτό από την ψυχροπολεμική ιστορική περίοδο που δεν ισχύει πια. Το άρθρο 4 ας πούμε του NPT θεωρείται κίνητρο. Έχει συμπεριληφθεί στη συνθήκη ως κίνητρο κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών που δεν έχουν ε, πυρηνικό οπλισμό. Τώρα όμως είναι εμπόδιο για την πυρηνική ασφάλεια. Γιατί θεωρείται δικαίωμα. Γιατί θεωρείται δικαίωμα ότι μπορεί κανείς να αναπτύξει όλες αυτές τις τεχνικές ενώ συγχρόνως έχουμε ένα εντελώς αναξιόπιστο και ανεπαρκές καθεστώς εγγυήσεων ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική μόνο για ειρηνικού σκοπού. Προσδοκούμε λοιπόν στην ε, μελλοντική διάσκεψη τη NPT και είναι πολύ ευτυχέ που μιλάμε για αφοπλισμό παρόλο την τελμάτωση στην οποία έχουμε περιέλθει επ' αυτού. Γιατί λέω τελμάτωση, γιατί προ το παρόν επικεντρωνόμαστε μόνο σε μέτρα διαχείριση τη υφιστάμενη κατάσταση ε, για την ε, που βασίζονται στην ειλικρίνεια ή μη των κρατών που έχουν πυρηνικά όπλα. Παρόλο λοιπόν που όλοι και περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι η ακολούθηση αυτή της ε, στρατηγική με το 2010 δεν θα οδηγήσει σε συμφωνία για ε, τις οποίες θα μπορέσουμε να εργαστούμε για τα επόμενα 10 χρόνια, παρόλα αυτά είναι ε, η κρατούσα άποψη. που κανείς δεν αμφισβητεί. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να την αμφισβητήσουμε, να την αναλύσουμε. Ο Χέλλη Κίσιντζερ σε ένα δημοσίευμά του ε, ανέφερε το θέμα του αφοπλισμού αλλά υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα και που ο ίδιος ανέφερε. Η θέση των είπα για τις δοκιμές, η θέση των ε, κρατών που έχουν πυρηνικά όπλα, η πυρηνική ασφάλεια, ε, η διάδοση σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη, ουράνιο-πλουτόνιο και η σταδιακή κατάργηση του εμπλουτισμένου ουρανίου σε μη στρατιωτικά προγράμματα. 13 βήματα είναι αυτά τα οποία προτείνουν ε, οι περισσότεροι και που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της διάσκεψης του 2000 ορισμένοι επίσης αναφέρουν ε, και την ολένα και μεγαλύτερη απειλή ιδιαίτερα μετά την 9η Σεπτεμβρίου της τρομοκρατίας. Προτάθηκαν τρία μέτρα, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν αναγνώριση του γεγονότος ότι τα θέματα ασφαλείας ε, για τα πυρηνικά δεν πληρούνται. Uh, and so they concluded, for example... Και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μείωση της εξάρτησης από τα πυρηνικά και τα σχετικά συστήματα, οι περισσότερες, οι περισσότερες περικοπές αυτά τα προγράμματα και η εξέταση των ε, περιφερειακών και τοπικών συγκρούσεων είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και το ίδιο το Wall Street Journal που βασίστηκε στις δηλώσεις ε, του ε, Πρόεδρου Ομπάμα έχει ασπαστεί τον στόχο ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Όχι διαχείριση και μείωση, κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι το ευκταίο αποτέλεσμα, διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να δράσουμε για να εφαρμόσουμε το όραμα που υπάρχει για ειρήνη και ασφάλεια. Ιδιαίτερα δε η Ένωση η προοπτική ενός ελεύθερου κόσμου από πυρηνικά είναι ρεαλιστική. Εξαρτάται όμως από τις σωστές δράσεις, στο μείγμα δράσεων. Αργά ή γρήγορα και καλύτερα γρήγορα παρά αργά θα πρέπει να γίνει αυτό χωρίς να χρειαστεί να υποστούμε τις συνέπειες μιας πυρηνικής καταστροφής. Υπάρχουν ανοιχτές πληγές από τον ψυχρό πόλεμο. Το αναγνωρίζω. Αλλά αν επικρατήσει αυτή η άποψη δεν θα έχουμε ασφάλεια δεν θα έχουμε κατάργηση πυρηνικών όπλων και ελεγχιστοποίηση της ε, από εκεί προερχόμενης απειλής. Το καθεστώς μη διάδοσης, όπως είπα, είναι ανεπαρκές, είναι αντιπαραγωγικό, ε, επιφέρει διακριτική μεταχείριση, ε, δεν εγγυάται την ασφάλεια και τον αφοπλισμό. Uh, most measures τα περισσότερα μέτρα που έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι επίμαχα. Είναι επίμαχα. Το πρόσθετο πρωτόκολλο για το οποίο έρχονται στην σειρά ετών, αλλά που πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ακόμα απειρχαιωμένο, ποτέ δεν ήταν σύγχρονο με άλλα λόγια που ο στόχο είχε να εμποδίσει το Ιράν να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου κτλ. είναι κάτι το οποίο ε, αποδείχτηκε αποτυχία η πρόοδος προς τον πυρηνικό αφοπλισμό μπορεί να μας βοηθήσει να επιλύσουμε κάποια από αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά θα πρέπει να συνοδευτούν με ένα σύνολο κανόνων και θεσμικών διευθετήσεων όλου του πυρηνικού καθεστώτος ευθύνε και της CIA και της NPT και όλων των ενδιαφερομένων το NPT το έχει αυτό κατά νου και στο θεματολόγιο του και εξετάζει σχετικά μέτρα και μέσα. Αν θέλουμε όμως να άρουμε αυτήν την πυρηνική δαμόκλεια σπάθη που ύπταται υπέρ των κεφαλών μας, που κρέμεται για την ακρίβεια υπέρ των κεφαλών μας, θα πρέπει να διαδραματίσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολύ σημαντικό και προδραστικό ρόλο είναι διάφορα τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Εγώ προτείνω τρεις πρακτικούς στόχους για τον αφοπλισμό που θα δημιουργήσουν ένα, μια πολιτική δυναμική και θα κινητοποιήσουν την κοινωνία. Είναι απλά και ορατά. Διότι ε, αν η κοινή γνώμη αν η κοινή γνώμη δεν απαιτήσει, δεν κατεβεί στον δρόμο να απαιτήσει τον αφοπλισμό, οι κυβερνήσεις ποτέ δεν θα το κάνουν από μόνες τους. Πρώτο βήμα να ξεκινήσει μια διαδικασία προς μια διάσκεψη για τα πυρηνικά όπλα που θα χαρτογραφήσει και θα πλαισιώσει τους στόχους για την σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Στην ε, NPT Review Conference του 2010 πολλά κράτη-μέλη θα ζητήσουν διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Ορισμένοι μπορεί να αναφέρουν ε, το σχέδιο του Μπανκιμούν 24 ε, Οκτωβρίου του 2008 πως πρώτο σημείο, ως βασικότερο σημείο είχε την ύπαρξη ενός νομικού νομοθετικού πλαισίου για την σταδιακή κατάργηση και απαγορευσή της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Άλλοι από πρακτική άποψη έθεσαν καταληκτική προθεσμία για την εκκίνηση διαπραγματεύσεων για μια τέτοια συνθήκη. Το 2020 έχει αναφερθεί μια τέτοια καταληκτική προθεσμία. Όπω και με τι συνθήκε για τα βιολογικά και χημικά όπλα, μια τέτοια συνθήκη για τα πυρηνικά θα κυριαρχούσε παλαιότερων νομοθετικών μέσων και θα ενδυνάμωνε το καθεστώ μη διάδοση και βεβαίως θα επικύρωνε όλα τα ψηφίσματα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας περιλαμβανομένων των 1887 και 1440. Θα είχαμε έτσι πολύ πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς και ελέγχους για την ε, περαιτέρω μη διάδοση των πυρητικών όπλων. Με τον στόχο αυτό μπορούμε να ασχοληθούμε με το πυρηνικό υλικό, με την διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και αυτών των εγκαταστάσεων που οδηγούν σε κατασκευή πυρηνικών όπλων. Έτσι θα έχουμε αφοπλισμό. Δεύτερο βήμα. Πριν την ε, διάσκεψη ως ένα μεταβατικό ενδεχομένως βήμα, όπως αναφέρει ο κ. Πασκάλ, να αναγνωρίσουμε ότι για χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Όχι να το αναγνωρίσουμε απλώς, αλλά και να το νομοθετήσουμε. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να απαγορεύσουμε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Όσο μειώνονται τα πυρηνικά οπλοστάσια, τόσο πιο σαφές θα καταστεί ότι δεν υπάρχει χώρος για νέες πολιτικές με βάση το πυρηνικό δόγμα και έτσι δεν θα δεχθούμε ούτε από ηθική, ούτε από νομική, ούτε από στρατιωτική ή πολιτική άποψη την χρήση αυτών των όπλων. Ούτε από μας, ούτε ε, όταν τα χρησιμοποιούν άλλοι. Και τρίτο, ένα κράτος μέλος που έχει πυρηνικά θα πρέπει να τα αποποιηθεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε κάποια βήματα προ αυτή την κατεύθυνση χωρί βεβαίω να τα ολοκληρώσει, χωρί να τα φτάσει μέχρι τέλου. Διότι παρέλυσε από τον φόβο ότι θα απομονωθεί. Ιδιαίτερα εφόσον θα άφηνε σε αυτή την περίπτωση μόνη τη την Γαλλία ω την μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο βεβαίω είναι ταμπού και αποκλείεται εξορισμού. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε αλλά και οι χώρε του ΝΑΤΟ του χρόνου θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να κινηθούν προ την αποπυρηνικοποίηση τη Ατλαντική Συμμαχία. Και πολλοί πιστεύουν ότι με την κατάργηση των πυρηνικών όπλων από το ευρωπαϊκό έδαφος θα κάνουμε ένα βήμα προ αυτή την κατεύθυνση. Αν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβουν ηγετικό ρόλο προ το στόχο αυτό, αν αποποιηθούν τα πυρηνικά όπλα, εάν δεχθούν ότι το πυρηνικό δόγμα είναι λάθος και ότι η κατοχή των πυρηνικών όπλων δεν αποτελεί ασφάλεια αλλά επαπειλή, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Εν κατακλείδη, δεν θα είναι εύκολο να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα, είναι όμως παντελώς ρεαλιστικό, απόλυτα ρεαλιστικό για να μην ξαναδούμε κι άλλα Ιράν, για να μην υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση και ενδεχομένως μια πυρηνική καταστροφή είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Πολλά από τα στοιχεία των 13 αυτών βημάτων, των 13 αυτών σταδίων είναι στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών ηγετών. Θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Εάν θέλουμε να μετακινήσουμε την ισορροπία προς μία αποπυρηνικοποίηση όμως, θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω πρακτικά βήματα για την ε, διάλυση των πυρηνικών οπλοστασίων και εγκαταστάσεων, για τον έλεγχο της διαδικασίας αυτής, για την αξιοπιστία της διαδικασίας ελέγχου, για την αποστρατικοποίηση της διεθνούς πολιτικής. Ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει να το κάνουμε, διότι γίνεται ολοένα και πιο ευρέως παραδεκτό ότι μία παγκοσμίω εφαρμοζόμενη πυρηνική συνθήκη είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο, τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να καλλιεργήσουμε. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά μεταβατικά μέτρα ούτω ώστε η απειλή και η χρήση των πυρηνικών όπλων να θεωρηθεί αθέμητη, παράνομη. Αυτό είναι ένα βήμα που απαιτεί τα εθνικά κοινοβούλια και τις εθνικές κυβερνήσεις να δηλώσουν ότι κατά την άποψή τους οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Η επίτευξη της κρίσιμης μάζας προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ζητούμενο για έναν πραγματικό αφοπλισμό. Οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις μας είναι πολύ ακόμα ε, διστακτικές πολύ επιφυλακτικές και θέλουν άλλος να δώσει το παράδειγμα. Δεν τολμούν να το κάνουν αυτές. Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών όμως και η κοινή γνώμη θα πρέπει να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση για να βρουν το κουράγιο οι πολιτικοί να λάβουν αυτές τις θαραλέε, ομολογώ αποφάσεις και να ετοιμάσουν έτσι το δρόμο των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια παγκόσμια συνθήκη από Τρει Τρεις πολύ σύντομες προτάσεις. Ένα, η Ένωση όπως και το 2000, να συντάξει ένα έγγραφο εργασίας που θα αποτελεί ένα συμπίλημα όλων των δηλώσεων των Ευρωπαίων ηθινόντων μέχρι το 2010 και που θα αποτελεί και που θα αποτελεί και μια έκκληση προς τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την διάσκεψη για την αποπυρηνικοποίηση. Δεύτερον, μια πανευρωπαϊκή διαδικασία διαβούλευσης και ερεύνης για το πώς θα αποπυρηνικοποιήσουμε τις στρατιωτικές, πολιτικές και πολιτικές ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. Με μη πυρηνικά όπλα δηλαδή να γίνονται αυτές οι πολιτικές αποτροπής αλλά και ασφαλείας. Δύναμη της ΚΕΠΑ και βεβαίως και τη συνθήκη της Λισαβόνος. Και τρίτον, να δημιουργηθεί η δυναμική για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους και τις κυβερνήσεις στο τέλος να προβούν στην θαραλέα δήλωση ότι θεωρούν, θεωρούν λέγω, ότι η οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Merci. Σας κατευχαριστώ κυρία Τζόνσον. Τώρα ο καθηγητής Μάσαλα. Και αμέσως μετά η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση, αλλά ήθελα να πω ότι οι τρεις ομιλητές που αναφέρθηκαν στη Σιμίδα συμφώνησαν λίγο πολύ. και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι έτσι η συζήτηση θα γίνει κάπως πιο αμφιλεγόμενη, γιατί ο, η Δόκτωρ Τζόνσον ή ο Δόκτωρ Τζόνσον ανέφερε ότι ο κύριος, ο τελικός στόχος είναι η πλήρης απαγόρευση. Το 2010 ξέρουμε ότι στο Παρίσι θα οργανωθεί μια τεράστια διάσκεψη όπου θα προσέλθουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και θα υποθεί ότι και το Global Zero είναι μια θεμητή επιλογή. Όλοι αυτό θέλουν τελικά. Γι' αυτό δεν θα ξανααναφέρω τα, τις πρακτικές συστάσεις που είπαν άλλοι και για να σεβαστώ και το χρόνο μου θα περιοριστώ στο ερώτημα που μου έθεσαν οι οργανωτές. Αν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε έναν κόσμο ελεύθερο πυρηνικών. Ένα ερώτημα που ποτέ δεν συζητιέται είναι όμως το εξής. Αν θα ήταν ευκταίο να υπάρξει κάποτε ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά. Αυτό που λέμε global zero. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ούτε ρεαλιστικό ούτε ευκταίο και θα αναφέρω τρία επιχειρήματα για το λόγο για τον οποίο δεν τον βρίσκω τέτοιο στόχο ρεαλιστικό και ένα επιχείρημα για το, κατά το οποίο δεν είναι και ευκταίο. Γιατί ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά θα είναι πολύ ασταθέστερος ενώ οι περιορισμένες πυρηνικές δυνάμεις θα μπορούσαν με πιο λογικό τρόπο να διαχειριστούν τα πράγματα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις σας λέω από την αρχή ότι με πληρώνει μεν η Γερμανία αλλά δεν εκπροσωπώ εδώ τις απόψεις της επίσημης Γερμανίας για το Global Zero που λένε. Και δεύτερον, πώς, πώς, και δεύτερον, προσωπικά είμαι υπέρ μιας μαζικής μείωσης Because I don't think that there is any strategic rationale for keeping more than 2000 αποθεμάτων πυρηνικών όπλων. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να επιστρέψουμε σε μια έννοια που είχε αναπτυχθεί το 70 και το 80 και που είναι πολύ υποσχόμενη για το μέλλον, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε μεν πυρηνικά όπλα αλλά όσο δυνατόν λιγότερα. Εγώ δεν είμαι ε, από τους πολεμοκαπήλους που ζητούν όλο και περισσότερα πυρηνικά όπλα. Απλώς θεωρώ ότι η κατάργησή τους δεν είναι ρεαλιστική ούτε και ευκταία. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα επιχειρήματα για τα οποία, με τα οποία εξηγώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να υπάρξει κόσμος χωρίς πυρηνικά. Πρώτον, οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ρωσία δεν θεωρούν αυτή την επιλογή τίποτε παραπάνω από μία απλή ρητορία. Δεν τη θεωρούν ρεαλιστική επιλογή. Πρόσφατες αποφάσεις του Πενταγώνου για τον εξυγχρονισμό των πυρηνικών καθώς και η απόφαση της Ρωσίας να χορηγήσει ακόμα ψηλότερα κονδύλια και για τακτικά πυρηνικά όπλα θα πρέπει να οδηγήσουν τους πολεμίους τους σε απορία. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ και ο Πρωθυπουργό Πούτιν και πολλοί στρατηγοί δήλωσαν ότι οι Ρώσοι δείχνουν ότι οι Ρώσοι δεν σκέφτονται καν την περίπτωση αυτή ούτε και σε 30 χρόνια γιατί θεωρούν τα πυρηνικά όπλα και την αποτροπή που αντιπροσωπεύουν αυτά ως ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής τους. εφόσον βέβαια ο στόχος είναι να αποτρέψουν τις υπόλοιπες χώρες από το να επιτεθούν στη Ρωσία και το ίδιο σκέφτονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρωσική πυρηνική πολιτική και η αμερικανική δεν δείχνουν καμία τάση έγκρισης της επιλογής αυτής του Global Zero. Άρα ο εξυγχρονισμός των πυρηνικών όπλων που, θα που έχουν αποφασίσει και θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια δεν πρόκειται να φτάσει να, τα μειώσει μέχρι το μηδέν. Και έπειτα είπε και ο προηγούμενος ομιλητής ότι η πρόταση αυτή για το Global Zero δεν εξαρτάται μόνο από τις Ηνωμένε Πολιτείες και τη Ρωσία. Πρέπει να συμφωνήσουν κι άλλοι. Και μέχρι τώρα οι περισσότερες υπόλοιπες πυρηνικές δυνάμεις είναι μάλλον χλιαρές για να μην πω τίποτα λιγότερο ως προς την επιλογή αυτή. Η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν απλό εξυγχρονισμό των πυρνικών. Η Ινδία, η Κίνα και άλλοι αυξάνουν τον αριθμό των πυρνικών τους κεφαλών. Και στο ΝΑΤΟ τελευταία συζητήθηκε η, μια νέα, η λεγόμενη νέα στρατηγική προσέγγιση ώστε να έχει μεν άλλο διαφορετικό ρόλο το ΝΑΤΟ αλλά όχι μηδενικό, ούτε μηδενική χρήση των, και διαχείριση των πυρηνικών. Αυτά θα τα ξαναδούν μέχρι το 11. Εφόσον λοιπόν δεν συμφωνούν όλες οι πυρηνικές δυνάμεις, δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι οι μεγαλύτερες από αυτές, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα συμφωνήσουν να ληφθούν μέτρα για την κατάργησή τους, αφού δεν θα τους ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Όσο για τη θέληση χωρών σαν τη Βόρεια Κορέα να καταργήσουν τα πυρηνικά ή του Ιράν να σταματήσει τις προσπάθειές του εμπλουτισμού δεν είναι επίσης ρεαλιστικές. Οι αντιδράσεις των υπολείπων πυρηνικών δυνάμεων δείχνουν ότι δεν υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός για τη μηδενική επιλογή. Άρα δεν είναι ρεαλιστική. Επίσης, αν το Ιράν πυρηνικοποιηθεί, τότε αναμένεται και άλλες χώρε της Μέσης Ανατολής και του Περσικού κόλπου, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, μπορεί να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο της πυρηνικοποίησης και όχι του, της κατάργησης των πυρηνικών. Τρίτον, ας υποθέσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πια πυρηνικά. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, αλλά η γνώση της παραγωγής τους υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει. Αφού όμως το τζίνι έχει βγει από το λιχνάρι εδώ και πολύ καιρό, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να μην εφαρμόσει τη γνώση, την τεχνολογία δηλαδή που θα διαθέτει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι χώρες ή άλλοι μη κρατικοί παράγοντες δεν θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή για να δημιουργήσουν, για να παραγάγουν νέες πυρηνικές κεφαλές. Και μάλιστα σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά ο πειρασμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Γιατί λόγω της τεράστιας καταστροφικής, του τεράστιου καταστροφικών δυνατοτήτων που έχει το όπλο αυτό, όλοι θα προσπαθήσουν να εξοπλιστούν περισσότερο από τους υπόλοιπους για να μπορούν να χτυπήσουν πρώτοι. Άρα, σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά θα είναι τεράστιες, τεράστιοι οι πειρασμοί. Λέω λοιπόν ότι η τεχνολογία υπάρχει και είναι γνωστή και θα αποτελέσει κίνητρο για άλλες χώρες ώστε να προσπαθήσουν και αυτές να παραγάγουν πυρηνικά. Γιατί λοιπόν ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά να θεωρούμε ότι δεν θα δημιουργήσει νέο ανταγωνισμό των εξοπλισμών από χώρες, κράτη ή και ομάδες μη κρατικές. Κατ' Αυτό δεν το έχουν σκεφτεί. Και φυσικά η μηδενική επιλογή, η Επιτροπή Υπερκατάργηση των Πυρηνικών ζητάει και ένα καθεστώς συνεχούς επαλήθευσης. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε μια χώρα που θα παράγει πυρηνικά ή που όπως το Ιράν θα παραβιάζει τις συνθήκες που έχει υπογράψει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι μηχανισμοί εξακρίβωση επαλήθευση επιτήρησης πρόκειται να δώσουν αποτέλεσμα. Και είπα ότι όχι μόνο χώρε, αλλά και μη κρατικοί παράγοντες θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να παραγάγουν πυρηνικά όπλα γιατί δεν μπορούμε να σβήσουμε τη γνώση της τεχνολογίας αυτής. Αυτά είναι τα κύρια επιχειρήματα, προσθέσω ένα. Εκείνοι που, ακόμη και οι χώρες που θα έχουν καταργήσει τα πυρηνικά τους, θα έχουν και αυτές την τεχνολογία και τη δυνατότητα όποτε θέλουν να τα ξαναπαραγάγουν. Άρα όποτε σημειώνεται μια κρίση θα ξαναρχίζει πυρηνικός ανταγωνισμός και οι μηχανισμοί των, της τελευταίας που διασφάλιζαν ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει πυρηνικός πόλεμος, οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα υπάρχουν πια. Άρα ο κόσμος θα γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος αν δεν υπάρχουν μεν τα πυρηνικά αλλά υπάρχει η τεχνολογία. Και αυτό με οδηγεί στο τελευταίο μου επιχείρημα κατά το οποίο δεν είναι ούτε καν ευκταίος ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά. Στην συζήτηση ούτε αυτό έχει ακόμη υποθεί και στην Ευρώπη έχει σχεδόν ξεχαστεί. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στην ιδέα ότι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα δεν χρειάζεται να, ότι κατά τις περιόδους αυτές δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την πυρηνική ενέργεια ή τα πυρηνικά όπλα. Και ότι δεν χρειάζεται πυρηνικό οπλοστάσιο, ότι είναι μάλιστα μη ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι τα στρατηγικά ή τακτικά πυρηνικά όπλα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ. Μπορεί να είναι σωστό το επιχείρημα αυτό, αλλά αγνοεί το γεγονός ότι η σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων αποτελούσε παράγωγο της, του γεγονότος ότι υπήρχαν τα πυρηνικά. Η κατάργηση τους σφαιρικά θα αυξανε τη δυνατότητα να σημειωθούν συμβατικοί πόλεμοι, ενώ η ύπαρξη των πυρηνικών ως απόπλων αποτροπής έδινε την εγγύηση της μακράς ειρήνης όπως είπε ο Τζον Λούις Γκάντης μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο εκμηδενισμός του θα σήμαινε ότι μπορεί να αυξηθούν εκ νέου οι συμβατικοί πόλεμοι και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά τα συμβατικά αποτρεπτικά όπλα. Έρχομαι λοιπόν στο συμπέρασμα. Προσπάθησα να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι ρεαλιστική η μηδενική επιλογή με τρία επιχειρήματα. Πρώτον ότι ο εξυγχρονισμός των οπλοστασίων σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο στεναροί πολέμοι των πυρηνικών δεν παίρνουν πολύ σοβαρά την ιδέα αυτή. Δεύτερον ότι οι ελάσσονες πυρηνικές δυνάμεις δεν πρόκειται να συμφωνήσουν και τρίτον ότι η κατάργηση των πυρηνικών οπλοστασίων δεν θα λύσει το κύριο πρόβλημα ότι υπάρχει η τεχνογνωσία για την παραγωγή των πυρηνικών. Και τέλος, σκεπτόμενος τι θα σήμαινε ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά, έδειξα ότι ένας τέτοιος κόσμος δεν θα κατέληγε σε περισσότερη ασφάλεια, αλλά στο αντίθετο. Άρα, η μηδενική επιλογή δεν είναι ούτε ρεαλιστική, ούτε ευκταία. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν πρέπει να πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειώνουμε τα υπάρχοντα πυρηνικά. Γιατί έτσι θα είχαμε τα ωφέλη των στόχων των ε, πολεμίων των πυρηνικών χωρίς όμως τις ελλείψεις. Ευχαριστώ κύριε Μασαλά οι τελευταίες ομιλίες, ο κύριος Μάσαλα και ο δόκτωρ Τζόνσον, ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες νομίζω και σας υπενθυμίζω ότι θα υπάρξει τώρα και συζήτηση και με τους πέντε, ίσως και μεταξύ σας, των πέντε. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα και ο ίδιος να θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτον, γενικά, αφού σας άκουσα και τους πέντε, ιδιαίτερα τους τρεις πρώτους τώρα, διαπιστώνω ότι σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε αναφέρει το 2005 στην προηγούμενη δηλαδή διάσκεψη της Σιμίδας ε, δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική πρόοδος. Έγιναν δηλώσεις της κυβέρνησης Ομπάμα, αλλά ως προς την ίδια τη διάδοση και την παραβίαση των κανόνων της συνθήκης από ορισμένα κράτη, όλα αυτά δεν αποτελούν καμία βελτίωση. Και άρα μπροστά σε αυτή την αυξανόμενη έλλειψη αξιοπιστίας της ημίδας και ιδιαίτερα τονίζω τον χαρακτήρα νότου-νότου της διάδοσης που είναι ενισχυτικός και πολιτικά και οικολογικά θα ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι μια απλή αναθεώρηση ή μεταρρύθμιση της συνθήκης αυτής αρκεί. Μήπως θα έπρεπε μια ολόκληρη καινούργια συνθήκη. Δεύτερο ερώτημα. Που ίσως να σας φανεί αφελές ιδιαίτερα εσάς, δόκτωρα Τζόνσον. Αναρωτιέμαι ειλικρινά, αναρωτιέμαι, κατά πόσον είναι ρεαλιστικά όσα δηλώνονται για τον αφοπλισμό. Γιατί σας ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω οι στόχοι, οι πολύ ευγενείς αυτοί οι στόχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση επί της τάσης των Βορειοκορεατών, των Ιρανών και των υπολείπων κρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων. που συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν πυρηνική τεχνολογία. Γιατί δεν μιλήσαμε για αυτήν τη διάδοση προς οργανώσεις, όχι μόνο προς κράτη. Τρίτο ερώτημα, συμπληρωματικό των άλλων. που το ανέφερε σύντομα όμως ο δόκτωρ Μάσολα, τι γνωρίζετε για την θέση των πυρηνικών όπλων στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ που πρόκειται σύντομα να αναθεωρήσει τη στρατηγική του. Τώρα έχουν ζητήσει το λόγο πολύ συνάδελφοι κυρία Λέζινγκ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευρύ το θέμα, πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μάσολα για αυτά που μας είπε. Συμφωνώ ότι έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Πολλοί δηλώνουν πολλά. Ως χριστουγεννιάτικες ευχές. Τα παραφορτώνουν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κι εγώ μπορώ να πω, Άγιε Βασίλη μου σε παρακαλώ κάνε τον κόσμο ειρηνικό, αλλά δεν πρόκειται αυτό να καταλήξει πουθενά. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μάσα, αλλά το ξαναλέω. Είμαι πολλά χρόνια ευρωβουλευτής και προσπαθώ πάντοτε να βλέπω τα πράγματα με ανθρώπινο και ρεαλιστικό τρόπο. Γιατί ξέρω ότι όποτε υπάρχει διαμάχη, ε, η διαμάχη έχει δύο μέρη. Όποτε έρχεται κάποιος δηλαδή να προσφύγει για διαμεσολάβηση, πάντοτε ο διαμεσολαβητής ζητάει να δει και τα δύο μέρη. Και τα δύο. Ε, το ίδιο πρόβλημα είναι. Το ίδιο πρόβλημα είναι και για τα πυρηνικά και για τα βλήματα. Μιλήσαμε για ρόλο της Ευρώπης, για αξιοπιστία, για τέτοια πράγματα. Αλλά αμέσως μετά μιλήσαμε για τα αλυτοκράτη αυτά, Βόρεια Κορέα, Ιράν και τέτοια και τα τρομερά πράγματα που κάνουν. Ξεχνάμε εδώ αυτά που μάθαμε στο σχολείο, τα βασικά δηλαδή. Την ιστορία ξεχνάμε. Δηλαδή η Κορέα ας πούμε, η Κορέα. Τι λέει η ιστορία της Κορέας. Ότι είχε συνεχώς διαμάχες. Και η σημερινή κατάσταση απορρέει από διαδικασίες πολιετής. Και η Δύση έχει αθετήσει υποσχέσεις της, όχι μόνο η Ανατολή. και η παράνοια της βορειοκορεατικής κυβέρνησης δεν είναι τελείως αβάσιμη. Υπήρξαν στρατιωτικές απειλές και από τη Δύση και η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να παρατήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα αν σεβαστούν τα βασικά της συμφέροντα. Αν την πιέσουμε όμως αν τις τριμώξουμε δεν θα δεχτεί να τα καταργήσει. Και αν θέλουμε να μην υπάρχουν πυρηνικά στην Κορεατική Χερσόνησο πρέπει να δοθούν εγγυήσει και να γίνουν υποχωρήσεις. Αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνευση. Πρέπει να ζητήσουμε συνεννόηση να υπάρξουν σύμφωνα μη επίθεσης, εγγυήσεις. Και πρέπει οι σειράξεις να στοχεύουμε στη μείωσή τους, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνουμε τις φιλικές προσεγγίσεις μια λογική προσέγγιση πάντα πετυχαίνει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν αποκλιμάκωση, αυτό είναι το θέμα. Όχι μόνο κόσμο χωρίς πυρηνικά, αυτό είναι πολύ απλοϊκό. Θέλουν ουσιαστική αποκλιμάκωση ή όχι. Ο στόχος είναι πάντοτε να υπάρξει μια φιλοδυτική κυβέρνηση, λένε, στη Βόρεια Κορέα και να διατηρηθεί η παρουσία των στρατευμάτων τους εκεί για να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι διατεθειμένες να προτείνουν ένα σύμφωνο μη επίθεσης και να μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία και είναι διατεθειμένες. Το ξαναλέω. Τέτοιες προτάσεις θα ήταν ενδιαφέρουσες και για τη Βόρεια Κορέα. Αλλιώς θα μας πούν δεν εξετάζεται τα συμφέροντά μας σοβαρά. Ναι, ξέρω ότι πρέπει να βιαστούμε πρώτα. Και κάτι ανάλογο ισχύει και για το Ιράν. Αυτό το έλεγα έτσι σαν παράδειγμα. Απλώς. Φίλεν Ντάγκ. Κύριε Γκαλτιέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές του πάνελ μας για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Υπήρχαν και διαφορές μεταξύ των τοποθετήσεων, αλλά όλοι συνεφώνησαν επί του ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το καθεστώς της μη διαδόσεως. Το πρώτο το οποίο λοιπόν θα ήθελα να πω το υπενθυμίσαν ήδη πολλοί από τους ομιλητές, δηλαδή μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών θεμελίων του καθεστώτος, μεταξύ των τριών πυλώνων του συστήματος που παγιώθηκε από τον ψυχροπολεμικό διπολισμό. Το σύστημα πλέον είναι πολυπολικό και όχι διπολικό. Αυτό εννοώ δηλαδή. Εξού και η σημασία των διαπραγματεύσεων start και συνέχεια αυτού. Follow-up δηλαδή. Και βεβαίω σημαντικός και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στον τομέα αυτό. Που θα πρέπει να, να αναγνωρίσει ότι είναι κομμάτι του προβλήματος. Του πυρηνικού προβλήματος εφόσον υπάρχουν πυρηνικές χώρες. Ή για να το πω καλύτερα, <laughs> χώρες με πυρηνική τεχνολογία και πυρηνικό οπλοστάσιο. Θα πρέπει λοιπόν να εξυπηρεθεί ένα κοινό παρανομαστής μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν πυρηνικά όπλα, αλλά και των διαφορετικών ευαισθησιών Ο κύριος Μέγερ είπε ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνος ήδη στην NPT μπορεί να γίνει αυτή η προσπάθεια εξέβρεση μια κοινή ευρωπαϊκής θέσεως. Και από πολιτική, αλλά και από θεσμική απόψεω. Και βεβαίω και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην προσπάθεια αυτή. Τώρα, θα είχα και κάποια ερωτήματα για μια σειρά θεμάτων. Πρώτα απ' όλα, εις ό,τι αφορά αυτά που είπε ο δόκτωρ Γκρό. για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε, νέο, σε νέα πυρηνική κούρσα, κούρσα εξοπλισμού, πυρηνικού εξοπλισμού σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. και ότι η κοινή γνώμη ανησυχεί στην Ιαπωνία, στην Τουρκία. Θα ήθελα τη γνώμη σας και για τη Βραζιλία. αλλά και για το ρόλο της Συρίας. Επίσης θα ήθελα την άποψη του δόκτωρος Γκραν λόγω της πρόσφατης επικαιρότητα και της δηλώσεως του Ιράν που βεβαίως θεωρήθηκε ως πολύ κακό από τους αναλυτές που όλα τα βλέπουν μαύρα βέβαια οι αναλυτές εννοώ. Για την όψιμη αποκάλυψη και δημοσίευση Θα ήθελα την άποψή σας για το τι μαγειρεύουν στο Ιράν. Πρόκειται όντως για ειρηνικό πρόγραμμα ή μήπω αυτό είναι απλώς ένα προπέτασμα καπνού. Και ποια είναι η πραγματική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει ανεξάρτητα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα μπορούσατε να επισέλθετε σε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκαλτιέρη. Κύριε Σανάκ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία που ελάβατε να συγκαλέσετε αυτή τη συνάντηση για ένα τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό ζήτημα. And so uh, I just uh, tabled question. Μόλις υπέβαλα στο Κοινοβούλιο μια προφορική ερώτηση, την οποία ενδεχομένω θα γνωρίζετε, την οποία ενέκρινε η ομάς μου, η πολιτική μου ομάς, η Άλντε με αυτό ακριβώς το περιεχόμενο, δηλαδή σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία της ομιλίας της κυρίας Ρεβέκας Τζόνσον. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε αμελητή προς την κατεύθυνση της κατάργησης των περιοτικών όπλων. Το ερώτημά μου μια νέα συνθήκη, ένα νέο σύμφωνο με, σε παγκόσμια κλίμακα για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Πώς θα γίνει. Και δεύτερον, πότε θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. About this issue. Είναι θέμα το οποίο συζητούμε επί δεκαετίες. Το σύμφωνο, η συνθήκη είναι η εκκίνηση μιας ευρύτερης διαδικασίας και ουχή ο τερματισμός της συνολικής προσπαθίας. Οι δηλώσεις Ομπάμα είναι πολύ καλές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αυτοί που λέγουν ότι αυτά δεν είναι ρεαλιστικά, δεν γίνονται, δεν εφαρμόζονται. Προς αυτούς θα ήθελα να πω το 1986 ή 87 στο Ρέικιαβικ ο κύριος Ρέιγκαν και ο κύριος Γκορμπατσόφ σχεδόν, σχεδόν συνεφώνησαν για την πλήρη κατάργηση των πυρηνικών όπλων εντός δεκαετίας. Το ξεχνούν αυτό πολύ είναι ένα επεισόδιο, της, ένα συμβάν σημαντικό της πρόσφατης ιστορίας. Αλλά εκεί, εις το μακρινό Then Gorbachev ο πρόεδρος Ρέικαν και ο πρόεδρος Γκορμπατσόφ σχεδόν, σχεδόν έφτασαν πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία λόγω της ανηθικότητος και της βλακείας αυτής των πυρηνικών όπλων δηλαδή. Πιστεύω ότι η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο, μπορεί να εγκρίνει ένα θεματολόγιο. Τα 13 αυτά βήματα. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κρίση του, ε, που έχουμε με το Ιράν ή τη Βόρεια Κορέα. πολλοί δεν κατανοούν. Ότι αλλάζει πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, τα πυρηνικά όπλα είναι νόμιμα σε αντίθεση με τα χημικά και τα βιολογικά. Μια χώρα που αποφασίζει λοιπόν να εφαρμόσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το κάνει. Όπως το έκανε η Βόρεια Κορέα. Η συνθήκη NPT είναι μια πολύ ασταθής και εύθραυστη ισορροπία που πολύ εύκολα καταστρατηγείται. Αποχωρεί κάποιος και τελείωσε η ιστορία. Δεν δεσμεύεται από τίποτα. Και από κανέναν. Αποχωρεί και με απόλυτα νόμιμο τρόπο φτιάχνει μια πυρηνική βόμβα. Ε, μια ατομική βόμβα εννοώ και μετά τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Μπαίνουμε δηλαδή στα πλαίσια ενός εφιαλτικού σεναρίου, αλυσιδωτών αντιδράσεων. Βγήκε η Βόρεια Κορέα, θα βγω και εγώ, μπορεί να πει μια άλλη χώρα. Βγήκε η Βόρεια Κορέα και εσύ, θα βγω και εγώ, λέει μια τρίτη χώρα. Και καταλαβαίνετε που το πάω. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την σταθερότητα παγκοσμίω, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην εντιμότητα των χωρών που έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Λυπούμε που το λέω, διότι η διεθνή κοινότητα δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα για να προλάβει αυτή την κατάσταση μόλις απαγορευθούν τα πυρηνικά όπλα, βεβαίως η Εθνική κοινότητα θα πρέπει να έχει έτοιμους τους απαραίτητους ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ε, βιωσιμότητα της απαγόρευσης. Δηλαδή που θα ελέγχουν πραγματικά ότι η Βόρεια Κορέα δεν κατασκευάζει ανεξέλεγκτα και ατιμωρητή πυρηνικά όπλα. Πρέπει να υπάρχει με άλλα λόγια ένα αξιόπιστο σύστημα κυρώσεων. Και όποιο λέει αξιόπιστο σύστημα κυρώσεων, λέει αποτελεσματικού ελέγχου. Δεν μπορεί να μιλά τα παιδιά για τα κακά του καπνού με ένα τσιγάρο αναμένο στο στόμα. Παραβολή είναι αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε στις χώρες που θεωρούμε εμείς κακές ότι μην έχετε πυρηνικά όπλα εσείς. Mm-hmm. Αλλά εμείς ε, είμαστε πιο έξυπνοι και έχουμε, ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτης με άλλα λόγια. Γι' αυτό δεν κατανοώ γιατί και πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Και όποιο παραβαίνει αυτή την απαγόρευση υφίσταται τι συνέπειε. Όπως γίνεται και σε άλλου τομεί, τον εμπορικό, το οικονομικό ή οποιονδήποτε άλλο. Κυρώσεις δηλαδή. Uh, Πρόκειται για έναν οικουμενικά εφαρμόσιμο μέτρο. Όποιος το παραβιάζει υφίσταται τις κυρώσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και ελπίζω ότι η προφορική μου ερώτηση που έχω ήδη υποβάλει και καταθέσει θα συμφωνηθεί και έτσι θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει στις εξελίξεις και να επηρεάσει προς τη θετική κατεύθυνση τα πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Με τη σειρά που έλαβαν το λόγο για να απαντήσουν με πιο εμπεριστατωμένο και εμβρυθή τρόπο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην ε, παρέμβαση του Μέζιγκαν. Ναι, ναι, σωστά, σωστά προφέρατε το όνομά μου, λέει η ενδιαφερόμενη. κυρία Μούζινγκ. Πολύ σωστά ε, είπατε ότι είμαστε ένα τμήμα της ιστορίας. Σε όλη τη συζήτηση και στην προσέγγιση ε, για το θέμα της ε, μη επεκτάσεως, μη διάδοσης ε, ασχοληθήκαμε με τα καθεστώτα και αυτό θέτει πολλά ερωτήματα διότι αναφερθήκατε στα παράνομα κράτη ε, rogue state που είναι μία ε, σωστή έκφραση για αυτό το σκεπτικό όπου διαπιστώνουμε ότι αν επικεντρωθούμε στο καθεστώς και θέλουμε το καθεστώς να αλλάξει σε αυτές τις χώρες, οι, ε, οι χώρες οι οποίες ε, κάθονται από την άλλη πλευρά του τραπεζιού δεν έχουν διέξοδο, διότι υπάρχει μία απειλή που δεν έχει σχέση με τα όπλα. Τα όπλα είναι απλώς ε, ένας τρόπος για να αυξηθεί η νομιμότητα του καθεστώτος και περί αυτού πρόκειται και και επ' αυτού επανέρχομαι στο Ιράκ διότι κατά τη δεκαετία του 90 μετά την απελευθέρωση του Ιράκ το Άνσκομ η, τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία ε, απέβλεπε στον αφοπλισμό και στην απομάκρυνση των πυρηνικών ε, ε, όπλων διαπίστωσαν ότι το Ιράκ είχε πρόγραμμα πυρηνικού εξοπλισμού και παραβίαζε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά ε, στη συνέχεια ε, προχώρησαν εις την απομάκρυνση του Σαντάμ Χουσέιμ και δεν υπήρχε λόγος να διατηρηθούν αυτά τα μέτρα. Οπότε και για το Ιράν πρέπει να διαχωρίσουμε πού είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ε, πυρηνικού προγράμματος και αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν εφόσον πρόκειται ε, για δύο γειτνιάζουσες χώρες προς ε, το Ιράν όπου απεμακρύνθη το καθεστώς στο Μέν Ιράκ με αμφισβητούμενες συνθήκες και στο Αφγανιστάν για σοβαρές και νόμιμες συνθήκες και διαδικασίες. Λοιπόν, όπως ε, αναφέρατε και την Κορέα και όπως αναφέρατε και το Ιράν, δεν θα δούμε καμία κίνηση, διότι το πρόβλημα δεν αναφέρεται πλέον στους πυρανικούς εξοπλισμούς, αλλά ε, απετέλεσε μόνο μία δικαιολογία για την ε, κατάργηση του συστήματος. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα ίσως να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα από τα θέματα και καταρχήν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εφέτος ουσιαστικά ε, είναι η πρώτη χρονιά μετά από το καθεστώς ε, και τη δίκηση Μπούς όπου ε, μετά από μία, ε, μία κυβέρνηση 8 ετή είμαστε σε μία περίοδο όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε ακολουθούν μία πολιτική πλέον ε, όπου θέλουν να διαχειριστούν την διάδοση και προσπαθούν, έχοντας προσπαθήσει στο παρελθόν να υποφεληθούν και να διαμορφώσουν την κατάσταση προς όφελός τους. Ε, τώρα όμως ε, η ρητορική έχει προχωρήσει χωρίς όμως να υπάρξει κάποια λύση στη Washington. Ε, υπάρχει μία στροφή, μία αλλαγή ως προς το σκεπτικό και ο, ο πρόεδρος Ομπάμα στην ομιλία του στην Πράγα ανακοίνωσε ότι οι ΙΠΑ θέλουν να ηγηθούν για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα όπλα, όχι γιατί ο κόσμος αυτός θα είναι καλύτερος, αλλά για ε, λόγους ε, αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή ότι μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατό να υπάρχει μια κοινωνία δύο τάξεων όσον αφορά τα πυρηνικά. Είναι το ίδιο σκεπτικό το οποίο είχε οδηγήσει τον, τον πρόεδρο Νίξον παλαιότερα να να προωθήσει την ε, κατάργηση των συμβατικών εξοπλισμών και όλα αυτά ε, τα μπορούμε να τα διαπιστώσουμε και ε, θα πρέπει να υπάρξει και μια συμφωνία για τα βιολογικά όπλα, για την απαγόρευση δηλαδή βιολογικών όπλων. Αυτά τα οποία αναφέραμε ούτως ή άλλως άπτονται στενά του, της τρομοκρατίας και ιδίως της πυρηνικής τρομοκρατίας και γι' αυτό θέλουμε να αποφύγουμε να διαδοθούν αυτά τα υλικά και να μπορούν να ελέγχονται. Το πόσο σοβαρή είναι αυτή η συνθήκη δεν αναφέρεται μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε και στις χώρες οι οποίες κατέχουν πυρηνικά όπλα αλλά και χώρες ε, ή συμμάχους που ε, δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Επ' αυτού υπάρχει μία ενδιαφέρουσα θέση της νέας γερμανικής κυβέρνησης η οποία ρητός έχει ταχθεί υπέρ ενός ε, αποπυρηνικοποιημένου κόσμου και η, η Γερμανία θέλει επίσης να αποφύγει να υπάρχουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα επί, γερμανικούς, ε, επί γερμανικού εδάφους. Δηλαδή ε, γι' αυτό και ανακοίνωσε η Γερμανία ότι θέλει να καταργήσει αυτούς τους οπλισμούς. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκρυφθεί. Και ένα άλλο βασικό θέμα ε, έχει σχέση με την τελευταία παρατήρηση την οποία άκουσα με πολύ ενδιαφέρον διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην παγκοσμιοποίηση έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα και τώρα βγαίνουμε από μία διοίκηση οκταετή ε, του Μπούς στην Αμερική και ό,τι ε, τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν είναι από το Δεκέμβριο του 2008 όταν ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή είχε στείλει μια επιστολή στον Μπαν με οκτώ σημεία τα οποία ε, ε, με μια εξαίρεση υπάρχουν σε όλα τα προηγούμενα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως άρα θεωρώ ότι αυτά δεν είναι επαρκή. Χρειάζεται μια πιο σαφής ανάπτυξη και αυτό αυτό δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας ε, για τη διεθνή διάσκεψη η οποία θα έχει μία αυστηρή μερίσια διάταξη αλλά θα πρέπει κανείς κάπως να αποστασιοποιηθεί από αυτό το πλαίσιο και να δημιουργήσει έναν ειδικό μηχανισμό διαβουλεύσεων που θα μπορέσει να συζητήσει τα θέματα αυτά για να διαμορφωθεί μια ίδια θέση. Ευχαριστώ ευχαριστώ για όλα αυτά τα θέματα και όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα θέματα τα οποία σημείωσα. Καταρχήν, αν πρέπει να αναδιατυπωθεί η TNP θα σας πω ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή ε, υπάρχει δυνατότητα όχι να θεωρηθεί η NTP, ε, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να υιοθετηθεί όπως έχει γίνει και στο παρελθόν το 1995 και κατά κάποιο τρόπο το 2000 ε, ένα πυρηνικό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία π.χ. να επικεντρωθεί επ' αυτού, να υπάρξει ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο θα μπορέσει να αποτελείται από δύο σελίδες και να μπορέσει να προχωρήσει. Να είναι δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο θα είναι σύντομο, σαφές και θα αποτελέσει ένα φύλλο πορείας για τα επόμενα έτη. Το δεύτερο θέμα είναι ότι θα ήθελα να επανέλθω στο ότι είπε η κυρία Λέζινγκ. Δηλαδή δεν έχουμε και εμείς ένα μέρος ευθύνης έναντι της Βορείου Κορέας ή του Ιράν ότι δεν έχουμε αντιδράσει θετικά σε σε ορισμένα σημεία. Και εδώ νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι εμείς πρέπει απλούστατα να αναγνωρίζουμε τα δικά μας λάθη, διότι η συζήτηση δεν είναι από πού ξεκινάει και πού τελειώνει το θέμα αυτό, αλλά στα δύο θέματα για την Βόρειο Κορέα με τον αντιδραστήρα, όπου ήθελε η Ευρώπη να προσφέρει τον αντιδραστήρα, αλλά όπου δεν σεβάστηκε τις ανηλυμένες υποχρεώσεις της η Κορέα επί 10 ε, χρόνια, όταν της ζητήθηκε να διαλύσει αυτές τις εγκαταστήσεις αρνήθηκε και μπλόκαρε η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και με το Ιράν επανειλημμένως παρεβίασε τις υποχρεώσεις του το κράτος αυτό. Ε, κανείς δεν τους αφισβητεί τη δυνατότητα να προωθήσουν ειρηνικά προγράμματα και αντιλαμβάνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, ούτως ή άλλως ε, αμφιλεγόμενες συνεργασίες μεταξύ της Ρωσίας και του Ιράν με εμπορικές ανταλλαγές, άρα το Ιράν έχει ειρηνική πρόσβαση για την την ατομική ενέργεια, αλλά αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να προχωρήσουν σε πυρηνικούς εξοπλισμούς και θα επανέλθω στο θέμα αυτό μετά. Ε, για να μην περιοριστούμε ε, σε ένα αγγλογερμανικό διάλογο για την κατάργηση των πυρηνικών ε, οπλισμών. Σαν Γάλλος θα ήθελα και εγώ να βάλω το λιχταράκι μου. Δηλαδή να πω ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρξει ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα και γι' αυτό θα ήθελα να πω ρητός ότι αν επανέλθουμε στον ε, κόσμο του 39 ή του 14 δεν είναι αυτόν στον οποίο προσβλέπω. Ε, αλλά εάν υπάρξει μία συλλογική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλείας οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά και θα πρέπει να αναλυφθούν πολύ ριζικές τομές για να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό. Δηλαδή ε, να διατυπωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνει αποδεκτό. Αλλά θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες ώστε όλα τα σενάρια, τα ανησυχητικά, τα οποία ανέφερε ο κύριος Μασάλα και με τα οποία συμφωνώ όσον αφορά τους κινδύνους. Δηλαδή να μην πρημοδοτήσουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν ζαβολιές, να μην ε, ε, ε, ε, πρημοδοτήσουμε τον τελευταίο κάτοχο, όλα αυτά τα θέματα όπου πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά για να προχωρήσουμε. Από αυτή την άποψη θα ήθελα να πω ότι αναφερθήκαμε πολύ στα βιολογικά και χημικά και στους χημικούς οπλισμούς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο απαγορεύσεως αλλά θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέλειες λύσεις. Πολλές χώρες δεν φέρονται σωστά και ε, οι χώρες αυτές θα πρέπει να αναδειχθούν. Υπάρχουν λοιπόν όρια ε, και, ε, και μέσα στα όρια αυτά ενεχόμαστε να υπάρχουν και αλλού πυρνικά όπλα. Όσον αφορά τη συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ξέρω τι μπορεί ε, να ε, προσκομίσει επικοδομητικά η συζήτηση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι ένα μέρος των πυρηνικών αυτών εγκαταστάσεων βρίσκονται στη Γαλλία και στην Αγγλία. Εφόσον λοιπόν έχουν τη μερίδα του λέοντος αυτές οι δύο χώρες μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αν όλες οι χώρες στον κόσμο ε, σεβαστούν αυτό που έκανε η Γαλλία και η Αγγλία, δηλαδή κυρώσουν την ε, συμφωνία για την απαγόρευση των δοκιμών, ε, σταματήσουν να παράγουν σχάσιμα υλικά. Θα έχουμε ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα για έναν πιο ασφαλή κόσμο και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Επίσης, θα πρέπει οι χώρες αυτές να συμβάλλουν στον αφοπλισμό με μονομερή μέτρα τα οποία οι δύο αυτές χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει μειώνοντας κατά 50% τους εξοπλισμούς τους, να υπάρχει ε, μεγαλύτερη διαφάνεια, να αποδείξουν ε, ότι μπορεί αυτό να γίνει από πλευράς διαφάνειας, να αποδείξουν επίσης ότι δεν πρόκειται να εξυγχρονιστούν ε, οι εξοπλισμοί τους και υπάρχει εκεί μία διάκριση μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας από τη μία πλευρά και της Κίνας από τις άλλη, η οποία αυξάνει τους εξοπλισμούς της ενώ η Γαλλία και η Αγγλία τους μειώνουν και άρα ακόμη ε, και αν μειωθούν ε, κάτω από τις χίλιες κεφαλές ε, οι εξοπλισμοί της Ρωσίας και της, των ΗΠΑ θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και τους υπολείπους. Και όσον αφορά την στρατηγική ε, ιδέα ε, περί ΝΑΤΟ. Είχα συμμετάσχει σε μία συζήτηση αυτούς τους τελευταίους μήνες σχετικά με ε, το πυρηνικό μέλλον της συμμαχίας και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχουν ορισμένες εκατοντάδες πυρηνικά όπλα. Ο ρωσικός στόχος όμως είναι 250 και νομίζω ότι για να υπάρξει μείωση των μεγάλων τακτικών ρωσικών εξοπλισμών γι' αυτό προωθεί τους δικούς της ε, εξοπλισμούς ε, η, η Ατλαντική Σημασία ε, για να υπάρξει ένας περιορισμός και των τακτικών οπλισμών στην Ευρώπη. Επίσης οι σύμμαχοι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις όσον αφορά τη στρατηγική λύση ε, συντηρητικά διότι καταρχήν υπάρχει η πίεση του ΝΑΤΟ που βοηθά τους συμμάχους και αν το ΝΑΤΟ κάποια στη ε, ε, ε, βασίζεται στις, στους πυρηνικούς οπλισμούς οι οποίοι θα πρέπει να καταργηθούν τότε θα πρέπει να αποπυρηνικοποιηθεί η πολιτική αμήνης. Άρα υπάρχει και μια τρίτη λύση, η οποία όμως είναι ίσως πρώιμη τώρα, και θα πρέπει ακόμη να αποφανθούν διάφορες άλλες χώρες προτού ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει. Αλλά και εκεί το ΝΑΤΟ όπως είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν ένα σημαντικό ρόλο διότι οι πυρηνικοί εξοπλισμοί οι ελάχιστοι ε, της Ατλαντικής Συμμασχίας ε, έχουν πολύ μικρότερη σημασία από ό,τι πριν από 20 χρόνια, διότι ε, στο, σε, πριν από μία δεκαετία είχε 9.000 ε, οπλισμούς στο ΝΑΤΟ και τώρα έχει μερικές εκατοντάδες. Ε, όσον αφορά τη Βραζιλία δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητική διότι ε, παρουσίασε τε, τους οπλισμούς του αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχεί στα πλαίσια μιας διάδοσης η οποία δεν επικτείνεται σημαντικά στην ε, Λατινική Αμερική. Όπως ε, ξέρετε η Παλαιστίνη έχει βομβαρδιστεί ε, από το Ισραήλ. Είδατε ότι κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε αλλά όλοι κατά βάθος ανακουφίστηκαν για να μην υπάρχει και ένας νέος πυρηνικός παίκτη στην περιοχή ιδίω γιατί αυτός ο, ο, ο παίκτη θα μπορέσει να υποφεληθεί από βοήθεια από την Βόρειο Κορέα. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση για το Ιράν δεν είναι μία συζήτηση ε, μεταξύ δυνάμεων που προσπαθήσουν να ε, πείσουν μία χώρα να μην ε, εμπλακεί σε πυρνικούς οπλισμούς, αλλά θεωρούν ότι είναι μία επικίνδυνη τοποθέτηση του Ιράν και γι' αυτό υπάρχουν και τα ψηφίσματα. Εγώ δεν ε, νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι κάποια μέρα θα υπάρξει ε, μία ε, μία ε, προσπάθεια του Ιράν ε, και καλυμμένα ε, και υπό αθέα, αθώα προσχήματα να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο θα είναι πολύ επικίνδυνο για να χρησιμοποιηθεί εις τους αντιδραστήρες. Δηλαδή ο στόχος των Ιρανών διαμφισβήτητα είναι ε, η δημιουργία οπλισμών και τίποτα άλλο. Και για να απαντήσω στο ερώτημα σας, εγώ πιστεύω ότι το καθεστώς του, της Τεχεράνης, το οποίο δεν διακινδυνεύει τώρα, διότι έχουμε δεχθεί ακόμη και την παρανομία των τελευταίων εκλογών και ε, το Ιράν χρειάζεται ε, αυτή την ε, κρίση παρόλο που οι Ηνωμένε Πολιτείες τους έτειναν το χέρι για να δημιουργήσουν μία κρίση που θα τους βοηθήσει να παραμείνουν στην αρχή. Όσον αφορά τις κυρώσεις, οι οποίες είναι δυνατές, υπάρχουν διάφορες κυρώσεις οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί από την ε, ε, διεθνή κοινότητα. Είναι μία ε, μείωση των παραδόσεων όπλων που θα δυσχεράνουν τη θέση. Βέβαια υπάρχουν χώρες οι οποίες κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία παραδείγματος χάρη με τις παραδόσεις αυτές των συμβατικών όπλων και υπάρχουν και οι πύραυλοι S-300. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο δεν επηρεάζει την επιβίωση του πληθυσμού είναι το θέμα ε, του ε, εξευγενισμένου πετρελαίου διότι στην περίπτωση του Ιράν ο που είναι μια χώρα που εισάγει τη βενζίνη ενώ εξάγει το ακάθαρτο πετρέλαιο μας δίνει την, ε, την ε, εικόνα της ε, θέσεως του καθεστώτος. Δηλαδή ότι οι επιλογές της κυβερνήσεως την αποδυναμώνουν και δεν την διευκολύνουν στο Ιράν. Ευχαριστώ. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολλά ενδιαφέροντα. Θα βασιστώ σε δύο και ίσως καλό θα ήταν να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση του κυρίου Ντονζόν. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια απλή αναθεώρηση το 2010. Εγώ συνήθως έπρεπε να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ενώ συνήθως ε, αναλαμβάνω να σχολιάζω το καθεστώς της μη διάθεσης από την πρώτη συνεδρίαση της NPT το 1994. Ε, υπάρχει λοιπόν η θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως πριν από τη διάσκεψη του 2000 που βοήθησε ε, να υπάρξει διαφάνεια και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα 13, 13 βήματα. Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά τα κράτη να προσπαθήσουν να επιτύχουν για το 2010 μια καλύτερη αναθεώρηση και να κοιτάξουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ημερήσια διάταξη η οποία ουσιαστικά αναφέρεται στη διαχείριση της διάδοσης των πυρηνικών εξοπλισμών. Από τη μακρά όμως πείρα η οποία έχει συγκεντρωθεί μπορεί κανείς να πει ότι είναι πράγματα που τα έχουμε δει και ξαναδεί. Déjà vu. Τα 13 βήματα είχαν, ε, ήταν το αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων και κατέληξαν σε μία συμφωνία το 2000 σαν μέρος της συζήτηση, αλλά στη συνέχεια απερίφθησαν, ανετράπησαν και λίγο πολύ ακυρώθηκαν. Οπότε ε, εδώ βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή ιδίω με την Προεδρία Ομπάμα και ε, λόγω ενός μείγματος συγκυριών. Δηλαδή, ε, άνθρωποι σαν τον Κίσιγκερ δεν προωθούν τον πυρηνικό αφοπλισμό γιατί γίναν καλύτεροι άνθρωποι από τόμος, αλλά διότι αντιλαμβάνονται ότι τα πυρηνικά όπλα ουσιαστικά είναι τα πιο ασταθή και απειλούν την ασφάλειά μας ως είτε προχωρούμε είτε όχι προς έναν πυρηνικό αφοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν το, 20, ε, το 2010 να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία και σε κάποιο κείμενο και να ε, καταρτήσουμε ε, ουσιαστικά θέματα κλειδιά των 13 βημάτων παρόλο που δεν συμφωνώ για το Ιράν, δεν συμφωνώ με αυτό που είπε ο Καμίζ ότι μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία μείον ενός, πλην ενός και πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαχωρίσουμε ε, τα προγράμματα προς τα εμπρός για στόχους, για βήματα προς, ε, την, ε, προς τον ποινικό αφοπλισμό, προς το στόχο που προσπαθούμε να επιτύχουμε με μία ανασκόπηση των θεμάτων που αφορούν το Ιράν παραδείγματος χάνει και όπου δεν θα χρειαστεί ομοφωνία ενώ για άλλα θέματα ίσως χρειαστεί ομοφωνία. Όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν για να δούμε πώς πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιο βασικό από όλα αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία συζητήσαμε και επί των οποίων ελπίζω θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Διότι η NPT έχει μία αδύναμη διαδικασία. Ξεκινήσαμε την αναθεώρηση το 1995 και τώρα έχουμε ε, περισσότερα προβλήματα από ό,τι προσόντα. Οπότε θα έπρεπε να έχουμε πιο σύντομες ετήσιες συναντήσεις όπου θα εξετάζουμε συγκεκριμένα προβλήματα και προκλήσεις ε, ε, συγκεκριμένα σε έναν πολύ ρευστό και γρήγορα ε, ε, τροποποιημένο κόσμο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε επί μίας βάσης και συμφωνώ με τον Καμίγ. Διότι αν θέλουμε να υπάρξει κατάργηση των πυρηνικών οπλισμών, εγώ δεν μίλησα για το Global Zero, ε, εδώ υπάρχει μία αίμονη ιδέα με αριθμούς, ενώ ουσιαστικά πρέπει να επικεντρωθούμε στην ασφάλεια και ε, να τοποθετήσουμε τη βάση επί της οποίας θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σιγά σιγά ενισχύοντας, οι μεν θα πηγαίνουν πιο γρήγορα, οι άλλοι πιο σιγά, αλλά για να υπάρχει μία ε, συνθήκη πυρηνικών εξοπλισμών θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να επιλύσετε όλα τα προβλήματα, εκ των οποίων πολλά ανέρχονται στην εποχή του ψυχρού πολέμου και ανέφερε ο κύριος Μασάλα, δηλαδή ε, την αστάθεια των κρίσεων, τον κίνδυνο, ο τρομοκρατίας ή τρομοκρατών που οι οποίοι θα μπορέσουν ε, να ε, βάλουν τα χέρια τους σε τέτοιους οπλισμούς και ε, αντιθέτως με τα βιολογικά χημικά όπλα τα οποία μπορέσαμε και απαγορεύσαμε θα θα πρέπει να ε, κοιτάξουμε να τα περιορίσουμε και αυτά, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου είτε ε, μία τρομοκρατική οργάνωση, είτε μία παράνομη ε, κυβέρνηση ε, προσπαθήσει να υποκλέψει, να αγοράσει κάποιο κατάλοιπο πυρηνικού όπλου πολιτικά να μην μπορέσει να υποφεληθεί γιατί θα υπάρχει μια κατάσταση όπου ολόκληρος ο κόσμος θα έχει μηχανισμούς συγκεκριμένα όχι μόνο ε, για να καταστήσει υπεύθυνο αυτόν ο οποίος εκφράζει την απειλή, να τον ε, ε, οδηγήσει στη Χάγη για να δικαστεί, αλλά ακόμη και τους προμηθευτές, ακόμη και τους επιστήμονες οι οποίοι θα συμβάλλουν ε, να μπορέσει να τους ε, προσαγάγει στην Χάγη για να δικαστούν ε, όπως έγινε με τον Αντάμ Χουσέι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι δεσπότης στη χώρα του, αλλά μπορεί τελικά να προσαχθεί σε κάποιο δικαστήριο διεθνές. Είναι εξελίξεις οι οποίες δεν θα προχωρήσουν ε, από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα μπορέσουν να γίνουν προόδοι εντός 10 ετών, εάν υπάρχει πολιτική θέληση διότι ορισμένες διαπραγματεύσεις πρόθυσαν ορισμένα θέματα και η συνθήκη θα μπορούσε να βοηθήσει να τοποθετηθούν οι βάσεις για να καταργηθούν τα υλικά τα οποία είναι ευαίσθητα για διάδοση και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα δούμε στην ε, πυρηνική αντιμετώπιση των ΗΠΑ αν όντως εννοούν αυτά που λένε ή απλώς ε, πρόκειται ε, για κουβέντες του αέρα. Πιστεύω ότι ε, οι κινήσεις που γίνουν ε, τώρα μας αποδεικνύουν ότι έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχουν πολύ πιο υπεύθυνοι ηγέτες από ό,τι πριν από 10-20 χρόνια διότι τη δεκαετία του 80 εμείς θέλαμε να καταργήσουμε τη συνθήκη της Βασοβία, το σύμφωνο της Βασοβίας και να καταρρίψουμε το τείχος ε, του Βερολίνου και ούτε ο Γκορμπατσόφ ούτε η Θάτσερ πίστευαν ότι ήταν ε, εφικτό ή επιθυμητό. Και τελικά όλοι αυτοί και από τις δύο πλευρές ε, του παραπετάσματος βοήθησαν να προχωρήσουμε και ε, να κατατάξουμε τα πυρηνικά όπλα, ε, να τα συνδέσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, όλες λοιπόν αυτές οι αφισβητήσεις οδήγησαν σε μια αλλαγή η οποία όταν συνέβη συνέβη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα είχε φανταστεί κανείς αν καθόταν απλώς σαν τον κύριο Μασάλα και προσπαθούσε να μας ε, διατυπώσει και να μας παρουσιάσει γιατί αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Δηλαδή οι θεωρητικοί ε, πίστευαν και αυτοί ότι αυτό ούτε μπορούσε ούτε έπρεπε να συμβεί. Και έτσι τελειώνουμε το Ιράν, διότι ναι. όταν έγραφα το έγγραφο αυτό για τους διερμηνείς, ε, με, μου τηλεφώνησε το CNN, το BBC, το Al Jazeera σχετικά με τις δηλώσεις του Αχμεντινετζάν για τις νέες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του ουρανίου και πιστεύω ότι όλα αυτά ε, είναι θριαμβολογίες διότι προσπαθούν απλώς να παρακολουθούν ακολουθήσουν, να επεξέλθουν της αποκαλύψεως μιας παράνομης εγκατάστασης και ε, της αλλαγής από τον ε, κύριο Ελμπαραντέη προς τον Ιαπωνέζο διάδοχό του διότι η, ε, η Ιαπωνία μπόρεσε και ανέπτυξε όλες τις ε, προόδους της πυρηνικής ε, τεχνολογίας ε, ειρηνικά και αυτό λέει το Ιράν ότι θέλει να επιτύχει. Αλλά νομίζω ότι ε, εάν πιέζουμε τον Αχμεντινετζάντ, το μόνο που θα κάνουμε είναι να τον προκαλούμε να πιέζει και αυτός εναντίον μας και δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μία εκτόνωση και απομάκρυνση από τα πυρηνικά όπλα και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουμε είναι εάν μειωθεί η αξία των πυρηνικών όπλων να πάψουν να θεωρούνται σαν ε, ένα σύμβολο ανδρισμού όπως ε, στην Ινδία δηλαδή δεν πρέπει να γελάμε με τέτοια παραδείγματα διότι δυστυχώς ε, τα πυρηνικά όπλα συνδυάζονται με κάποια κάποια προβολή και σαν Ευρωπαίοι πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες του πυρνικού αφοπλισμού και να τα αποδεσμεύσουμε από την ιδέα της μεγάλης κυριαρχίας την οποία ούτως ή στην οποία ούτως ή άλλως είναι ακόμη προσελωμένες χώρες σαν την Αγγλία και την Γαλλία. Εγώ θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, όσον αφορά την δικιά σας ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, εάν η επεξεργασία αρκεί ή αν χρειάζεται μία νέα διαμόρφωση. Ουσιαστικά πιστεύω χρειάζεται μία νέα διαμόρφωση, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρά μόνο με την αναμόρφωση ιστορικά. Η ε, πρόκειτο ε, για έναν συνδυασμό μεταξύ πυρηνικών και μη πυρηνικών πτυχών και για την δικτακτορία των πυρηνικών έναντι των μη ε, πυρηνικών ε, κατεχόντων. Ε, αυτό το, ε, αυτοί οι συνθήκες δεν υφίστανται πλέον και πιστεύω ότι όσον αφορά τα εσωτερικά προβλήματα είχαμε και την Αμερικανική πολιτική ε, σε σχέση με την Ινδία ε, που οδήγησε στη δημιουργία νέων προβλημάτων αντί την εκτόνωση των προηγουμένων. Όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις της κυρίας Λόζινγκ η οποία έφυγε εντωμεταξύ νομίζω ότι όταν κοιτάμε την Κορέα και το Ιράν δεν ε, πρέπει να ασχολούμεθα μόνο με το άρθρο 6 της NPT αλλά και με την ε, ε, τοπική περιφερειακή θέση. Δηλαδή η θέση του Ιράν και της Βορείου Κορέας οφείλεται στην περιφερειακή τους θέση και τη σχέση τους με τους ατομικούς οπλισμούς και λιγότερο με τις ανεπαρκή ε, ε, τον ανεπαρκή σεβασμό των υποχρεώσεων των μεγάλων δυνάμεων έναντι της NPT. Και το τελευταίο θέμα σχετικά με τον ε, κύριο Αυλάκη, Σωστά είπατε ότι τότε θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να σκεφτούν πώς θα πρέπει να διατυπώσουν κυρώσεις για να υπάρξει ένας αφοπλισμένος κόσμος αλλά ε, τότε ε, ε, πώς, ποιος θα είναι ε, μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας διότι η νομιμοποίηση των πέντε δυνάμεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οφείλεται στο, στην κατοχή τους πυρηνικών όπλων. Ε, αυτό επιτρέπει στις χώρες αυτές να έχουν ε, βέτο διότι διαφορετικά θα χάσουν την νομιμοποίηση την οποία τους, την οποία τους κατηγορούμε τώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η λύση δεν είναι εφικτή. Και όπως είπε και η κυρία Τζόνσον, ε, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το όραμα, όραμα του ενός ή του άλλου. Το θέμα είναι εάν ε, είναι ε, μία κατάσταση επικίνδυνη, αν χρειάζεται ένα αποτρεπτικό μέσο για να μπορέσουμε να χαίρουμε αυτού του καθεστώτος ειρήνης και ασφαλείας που υπάρχει από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πονέμου. Δεν θέλω να αναφερθώ πέρα περαιτέρω, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο πιο ρεαλιστικός με την στάση που ακολουθεί. Μήπως κάποιος θέλει ακόμη να αντιδράσει στη, στα τελευταία σχόλια. Κύριε Αρλάκη, σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά δεν θα υπάρχει Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο αποτελείται από τις πυρηνικές δυνάμεις. Δεύτερον, φυσικά θα υπάρχει μια συνθήκη όπου βάσει της οποίας δεν θα τα διαχειρίζεται όλα το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά ένα πιο διευρυμένο, θα υπάρχει ένα πιο διευρυμένο σύνθημα εφαρμογής κυρώσεων, ένα άλλο καθεστώς δηλαδή επίσημης απαγόρευσης. Τα πυρηνικά όπλα θα είναι παράνομα και θα είναι παρανομία, έγκλημα να χρησιμοποιούνται. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα δικαστήριο, δεν χρειάζεται Συμβούλιο Ασφαλείας. Επομένως δεν είναι σωστή αντίρρηση αυτή που είπατε. Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε να μείνουν τα πράγματα όπως είναι και να έχουμε προβλήματα με οποιαδήποτε Ιράν κάθε μήνα, τότε όντως θα καταλήξουμε σε ανταγωνισμό εξοπλισμών, αλλά νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό και απλούστερο θα ήταν να πούμε στο Ιράν απαγορεύονται τα πυρηνικά όπλα, γι' αυτό δεν μπορείτε να τα έχετε. Είναι κατά της διεθνούς νομοθεσίας. Αυτό είναι επιχείρημα. Αλλιώς τι θα πούν οι Ιράνοι, θα πούν γιατί εμείς. Εσείς μας το απαγορεύετε γιατί είστε εναντίον μας, είστε αντιμουσουλμάνοι, και είναι και αυτό σοβαρό επιχείρημα. Και το δικό μου επιχείρημα θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε παντού και στην Κορέα και παντού. Και σε χώρες που αναμένουν να δουν τι θα κάνει το Ιράν για να χρησιμοποιήσουν τα ίδια. Αυτά είναι φιαλτικά σενάρια. Ούτε είναι σωστό ότι έχετε 181 χώρες όπως είπατε κατά του Ιράν. Η Βραζιλία εμπλουτίζει ουράνιος όπως το Ιράν. Και όμως έχει καλές σχέσεις και έχει καλές σχέσεις με το Ιράν γιατί καταλαβαίνουν τους λόγους για τους οποίους το κάνουν και οι δύο. Και άλλες χώρες στον κατάλογο της Διεθνούς ε, Υπηρεσίας Ατομικής Ενεργείας συμπεριλαμβάνονται. Δεν είναι οι μόνες αυτές. Λοιπόν, αν διατηρήσουμε ένα σύστημα όπως έχει, που είναι δομικά, που έχει δομική έλλειψη ισορροπίας, δεν θα καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά μέσω της ε, σημείνας. Γιατί πρέπει ριζικά να φύγουμε από την ΣΜΔ. Αλλιώς θα συνεχίσουν τα πράγματα για τα επόμενα 30 χρόνια όσοι έχουν αυτό είναι το επιχείρημα υπέρ μια τελείω νέα συνθήκη που να βασίζεται στην απαγόρευση και την οποία να έχουν εγκρίνει οι περισσότερες χώρες. Έτσι θα είναι πολύ πιο ισχυρή. Εγώ δεν πιστεύω ότι πράγματι το Ιράν είναι το κύριο πρόβλημα. Πιστεύω ότι οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη είναι ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος. Το Πακιστάν είναι πολύ πιο επικίνδυνο. πολλούς λόγους από κάθε άποψη είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το Ιράν. Διότι το Ιράν παίζει ένα εσωτερικό παιχνίδι και περιφερειακό. Πολύ παρόμοιο με του Ιράν και του Σαντάμ. Τραβάνε το σκηνή μέχρι στην περίπτωση του, όπως στην περίπτωση του Σαντάμ να σπάσει. Αλλά το Πακιστάν είναι άλλο θέμα. Μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνος παράγοντας. αν δεν αλλάξουμε ριζικά τα πράγματα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Για να δούμε τι κάνει το Ισραήλ, κάτι ανάλογο πολύ πιο κρυφά βέβαια. Αν πούμε σε όλους αυτούς, α, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, είναι έγκλημα και με αυτό συμφωνούν οι περισσότερες χώρες. Τότε θα τους βάλουμε σε πολύ δυσκολότερη θέση, γιατί η βασική κύρωση είναι το ταμπού να αντικατασταθεί με πλήρη απαγόρευση. Μόνο έτσι θα υπάρξει το σθένος που ζητήσατε και εσείς ο ίδιος. Ευχαριστούμε. Για να τελειώνουμε τώρα. Μήπως κανένας εμπειρογνώμων θέλει να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο. Για πολύ λίγο χρόνο βέβαια. Αν θέλετε ορίστε ορίστε. Ο Κάμιλος. Ε, αυτό το θέμα του Ιράν και τις θέσεις του διεθνώς. Στην IAEA e τελευταία, τρεις χώρες επί 40 εκφράστηκαν σαφώς υπέρ του Ιράν. Η Βενεζουέλα, η Κούβα, του Κάστρο ή των αδελφών Κάστρο και η Μαλαισία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα, καμία διεθνή στάση υποστήριξης του Ιράν. Βέβαια σωστά είπατε ότι δεν υπάρχει και ομοφωνία, αλλά λίγες χώρες υποστηρίζουν το Ιράν και αυτές είναι περιθωριακές στη διεθνή σκηνή. Δεν πρέπει να βάζουμε στο ίδιο τσβάλι ε, το Ιράν και την Ιαπωνία. Αυτό είναι προσβολή για την τελευταία η Ιαπωνία θεωρεί ότι υφίσταται πολύ περισσότερους διεθνείς ελέγχους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί έχουν περισσότερα πυρηνικά βέβαια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι στο Ιράν εδώ και 40 χρόνια. Και όλο το Ιαπωνικό πρόγραμμα βασίζεται σε αυτό το θέμα του διεθνούς ελέγχου, συνεχούς διεθνούς ελέγχου, μα όχι, εγώ μίλησα για τη Βραζιλία, όχι για την Ιαπωνία. Βραζιλία. Μήπως η μετάφραση είπε η Ιαπωνία. Όχι, εγώ μιλάω για την Ιαπωνία, δεν είπα ότι εσείς το αναφέρατε. Γιατί είπατε ότι το Ιράν ακολουθεί το Ιαπωνικό πρότυπο, κάποιος είπε. Και τέλος, για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ιστορικά δεν αποτελούνταν μόνο από πυρηνικές δυνάμεις, Βέβαια έτσι έτυχε τα πέντε μόνιμα μέλη να είναι και πυρηνικές δυνάμεις. Αλλά η Κίνα όταν ήταν ακόμη το Ταϊβάν στο ΝοΙΕ δεν ήταν πυρηνική δύναμη κτλ. Το να είναι κανείς πυρηνική δύναμη δεν σημαίνει ότι αυτομάτως έχει και θέσεις μόνιμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. οι μη πυρηνικές χώρες που σέβονται τις δεσμεύσεις τους όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία. Είναι κάτι πολύ σοβαρότερο. Είπα να μην βάζουμε στο ίδιο τσεβάλι την Ινδία, το Πακιστάν, το Ισραήλ και άλλα. Ναι υπάρχουν ανησυχίε για όλες αυτές τις χώρες και για το Πακιστάν ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι στην ίδια κατηγορία διότι, διότι διότι λέγω εδώ και 40 χρόνια αφήνουν ανοιχτή αυτή την πυρηνική επιλογή. Μπορεί κανείς να είναι ταχθεί κατά, να ζητήσει αφοπλισμό της χώρας, αλλά πάντως δεν έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ιδίως όταν είμαστε Ευρωπαίοι και άρα υπέρ της πολυπλευρικότητος. Εγώ ανέφερα ότι το Ιράν αναφέρει το ιαπωνικό μοντέλο, το ιαπωνικό παράδειγμα. Δεν είπε κανείς προς Θεού ότι, η Ιαπωνία ε, ε, ακολουθεί ε, το Ιράν και ότι θέλει να έχει πυρονικό οπλοστάσιο. Εγώ ομιλώ την Ιαπωνική, έχω επισκεφθεί τη χώρα, είμαι σε επαφή με τις Ιαπωνικές αρχές και υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει η δυνατότητα ενδεχομένως εάν οι πολιτικοί αλλάξουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Ιράν αναφέρεται στην Ιαπωνία συνέχεια. Λέει εμείς και η Ιαπωνία καμία διαφορά. Γιατί ελέγχετε εμάς και δεν ελέγχετε την Ιαπωνία το ίδιο. Αυτό λέει το Ιράν. Και είπα ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ενδυνάμει πρόβλημα. Αλλά αυτό που πραγματικά ήθελα να πω ήταν να απαντήσω στον κύριο Μασάλα που έθεσε πάλι αυτό το ζήτημα. Ότι αν δεν είχαμε πυρηνικά όπλα θα ήμασταν στην κατάσταση, θα περιερχόμεθα στην κατάσταση προ 45 και ότι η πυρηνική αποτροπή είναι αυτό που κράτησε την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη. Αναγνωρίζω ότι έχει πέρασει αυτό το επιχείρημα. Δεν αληθεύει, πιστεύω όμως. Ως επιστήμον γνωρίζω ότι δεν μπορεί κανείς να κοιτάξει το αποτέλεσμα και εξ αυτού να μαντέψει το λόγο. Όχι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα επιστημονικός πως ομιλώντας. Εγώ είχα την ευκαιρία να φάγω πρωινό με τον Ρόμπερτ Μακναμάρα και όλοι με ρωτούσαν αυτό το ερώτημα. Τα πυρηνικά μας διασφάλισαν την ειρήνη τα τελευταία χρόνια και μου είπε ο κ. Μακναμάρα δεν είναι αυτή η σωστή ερώτηση. Η σωστή ερώτηση είναι απέτρεψαν τη Σοβιετική Ένωση. Okay, Ωραία λοιπόν. Λέω τότε στον κύριο Μακναμάρα απέτρεψαν τη Ρωσία. Τη Σοβιετική Ένωση. Και είπε όχι. Όχι, όχι είπε την πρόθεση ουδής δύναται αποτρέψει, απήντησε ο κύριος Μακναμάρα. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βεβαίως δεν έγινε τίποτα κακό, αλλά την πρόθεση δεν μπορούμε να αποτρέψουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι οικασίες. Η Σοβιετική Ένωση είχε παγιώσει τη σφαίρα επιρροής της αλλά ποτέ καθ' τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν είχε την πρόθεση να εισβάλλει στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχτισε και τον τοίχο του Βερολίνου. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η Σοβιετική Ένωση ήταν να εισβάλλει στη Γερμανία.